Συνάδελφοι, καλώς ορίσατε συνεδρίαση της Επιτροπής μας, Επιτροπής ε, των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των Δύο Φύλων. Είναι η πρώτη μας ε, συνεδρίαση το 2010 και ελπίζω να στεφθεί με επιτυχία το 2010 για όλους τους συναδέλφους και για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην έναρξη των δραστηριοτήτων μας για το 2010 και στη σημερινή μας συνεδρίαση. Πρώτο σημείο είναι η έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Υπάρχουν τροπολογίες, όχι δεν έχω λάβει κάτι, οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σημείο 2 προηγούμενης συνεδρίασης που έλαβε χώρα στις 30 Νοεμβρίου του 2009. Δεν έχω λάβει καμία τροπολογία, καμία ένσταση. Και αν δεν προκύψει κάτι μέχρι το πέρας της σημερινής μας συνεδρίασης, θα εγκριθούν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το σημείο σήμερα. Περνούμε απευθείας στο σημείο 4. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας την κυρία Μπιμπιάνα Άιντο Αλμάγκρο. Παραφθύρω το όνομά σας κατά πάσα πιθανότητα. Είστε Υπουργό Ισότητα των Φίλων τη Ισπανία, τη χώρα τη ε, Προεδρία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να διαβιβάσετε και τις ευχαριστήσεις μας προς την Ισπανική Προεδρία για, την, ε, για ένα ταξίδι που έκανε ένα κλιμάκιο της Επιτροπής μας ε, στην Ισπανία. Πολύ ευχάριστη επίσκεψη και δράτω με της για να σας πω ότι χαιρόμαστε στην Επιτροπή μας που βλέπουμε ότι έχετε αναδείξει σε προτεραιότητα στο πρόγραμμά σας την ε, ισότητα των δύο φύλων και πιο συγκεκριμένα την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ας μένω σας καλωσορίζουμε λοιπόν από τον Απρίλιο του 2008 διατελείται υπουργό τη Ισότητα των Φύλων από την ίδρυση του ομώνυμου Υπουργείου δηλαδή. Καλώς ορίσατε. Και περιμένουμε με ανυπομονησία την ενημέρωσή σας και ε, τις επόμενες ευκαιρίες που θα έχουμε να συζητήσουμε τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή για την παρουσία μου, στην, παρουσία μου αυτή στην Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ισότητας των Ευκαιριών, σε αυτό το κοινό οίκο της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας για να σας εξηγήσω τους στόχους της εκπεριτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου σε θέματα ισότητας. Θα ήθελα καταρχήν ως Ευρωπαία Πολίτης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι έρχομαι εδώ σε ένα κοινοβούλιο με περισσότερες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις και στον έλεγχο της διακυβέρνησης Ένωσης. Η ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων είναι μια διάσυστη απόδειξη της πολιτικής οριμότητας του ευρωπαϊκού σχεδίου. Μια οριμότητα που αποτυπώνεται σε μια πιο δημοκρατική και υπεύθυνη έννοια μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας όπου η ιδέα της περισσότερης Ευρώπης ε, βρήκε το δρόμο της μετά από πολλές δυσκολίες και περιπέτειες, όπως συμβαίνει με όλα τα μεγαλεπίβολα συλλογικά σχέδια. Θα ήθελα λοιπόν να σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό γιατί είστε εκπρόσωποι των ε, πολιτών ε, της Ένωσης, ανδρών και γυναικών. Στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού, κυρίες και κύριοι, η Ισπανία θα αναλάβει με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα για τέταρτη φορά την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακολουθήσουν η Βελγική και η Ουγγρική Προεδρία. Με τι χώρε αυτέ συνεργαζόμαστε στενά εντό του νέου συστηματο του τριο για να εξασφαλίσουμε συνέχεια, σταθερότητα και συνοχή στο σχέδιο που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Ε, η Προεδρία μας είναι μια Προεδρία προόδου πολιτικών προτάσεων και πρωτοβουλειών, μια προεδρία συνεργασία και αφοσίωση με τα θεσμικά όργανα τη Ένωση και με τα νέα αξιώματα του μόνιμου Προέδρου του Συμβουλίου και τη ΥΠΑ τη Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική. Θα υποβάλουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των τριών χωρών του Τρίου για τους επόμενους 18 μήνες, ένα κοινό πρόγραμμα που θα παραμείνει πιστό στις ιδρυτικές αρχές της Ένωσης, ε, μία από τις οποίες είναι η ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μία ισότητα που θεωρούμε ως οριζόντιο και κοινό στοιχείο όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή την άποψη θα κάνω ιδιαίτερη μνήα στον πρωταρχικό στόχο της Ισπανικής Προεδρίας στην Ένωση την ανάκαμψη της οικονομίας και την ε, αναζωογόνηση της απασχόλησης. Κυρίε και κύριοι, εφιστάμεθα ακόμη τι επιπτώσει τη σοβαρότερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ζήσαμε σε παγκόσμιο κλίμακα τα τελευταία 60 χρόνια και μάλιστα με ιδιαίτερε συνέπειε στην απασχόληση. Παράλληλα, η Ευρώπη έχει εντρυφήσει στον προσδιορισμό ενό νέου αναπτυξιακού οικονομικού μοντέλου για την επόμενη δεκαετία μετά την εκπνοή τη στρατηγική τη Λισαβόνα, που οι στόχοι τη δυστυχώ δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρω μια εργασία που θα γίνει με βάση τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία συνεργαζόμαστε στενά σε ό,τι αφορά την αποδοχή και την ενσωμάτωση των προτάσεων των κρατών μελών. Είμαστε επιπισμένοι ότι σημείο φετηρία τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική θα πρέπει να είναι η βιωσιμότητα, η αηφορία, δηλαδή η ικανότητα ικανοποίηση των παρουσών αναγκών, χωρί όμω να διακυβεύσουμε τις απαιτήσει του μέλλοντος. Και η φορεία σε τρεις ε, τομείς. Στον τομέα της οικονομίας, εκεί θα δώσουμε έμφαση στους τομείς της γνώσης και της ε, καινοτομίας. Στο περιβάλλον, που θα δώσουμε έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θα ενταχθούν στην, καταπολέμηση, στην προσπάθεια καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών και κοινωνική εφορία και βιωσιμότητα και θα φέρουμε τον πολίτη στο επίκεντρο της πολιτικής δράσης. Θα γίνει ο πολίτης ο άξονας της πολιτικής δράσης. Θα είναι ο απότερος στόχος της οικονομίας απέναντι σε άλλες θεωρίες και δόγματα που μας οδήγησαν στην οικονομική και χρηματοπιστωτική καταστροφή την οποία ακόμη βιώνουμε. Διανύουμε μια κρίσιμη στιγμή και θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια σημαντική καμπή της κοινωνίας μας προς ένα πιο ε, λογικό, δίκαιο, αλληλέγγυο και αποτελεσματικό μοντέλο. Και από την άποψη αυτή θα πρέπει να υπολογίζουμε στις αρχές και στις πολιτικές της ισότητας. Γι' αυτό ένα σημαντικό στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020 είναι η πλήρης ένταξη και σωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας, επίσης όρις με τους άνδρες. Αυτό θα είναι απαραίτητο στοιχείο για την εδραίωση της οικονομικής ανάπτυξης. Κάτι που περιλαμβάνεται άλλωστε στα συμπεράσματα της ε, Σουηδικής Προεδρίας και εγκρίθηκαν στο τελευταίο Συμβούλιο του 2009. Η στρατηγική της Λισαβόνας είχε μεταξύ των στόχων της τη ισότητα ανδρών και γυναικών, καθώς και την κοινωνική ένταξη. Φτάσαμε το 2010, χωρίς όμως να έχουμε υλοποιήσει πλήρως τους στόχους αυτού. αυτούς. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει να υποτιμούμε το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα, ούτε και την κατεύθυνση που ορίσαμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πλήρη ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασία, αλλά και σε όλου του τομεί τη ζωή. Γιατί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι μόνο δίκαιη από την άποψη των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά είναι και αποδοτική από οικονομική άποψη. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρέπει να ενισχύσουμε όλε τι πολιτικέ που στόχο έχουν την προαγωγή τη ισότητας αυτή. Η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν μπορεί να στερηθεί την ικανότητα, την ευφυΐα και το ανθρώπινο κεφάλαιο του μισού της πληθυσμού, που είναι οι γυναίκες. Γι' αυτό και όλες μας οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στον εντοπισμό και τη διόρθωση των εμποδίων που πολλές φορές παρακολύουν και άλλες φορές δυσκολεύουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, επίσης όρις με τους άνδρες. Το πρώτο αυτό εμπόδιο είναι η πρόσβαση και η παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων γιατί οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη φροντίδα των εξαρτημένων ανθρώπων, δηλαδή των ή ηλικιωμένων στην οικογένεια ή και των παιδιών. Αυτό όμω δεν είναι αποκλειστικό πρόβλημα των γυναικών. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε ενάψματα για να γίνει ένα πιο δίκαιο καταμερισμό ε, του χρόνου φροντίδα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ώστε να εναρμονίσουμε τη διαθεσιμότητα και των δύο στην εργασία. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να κάνουμε ένα ακόμη βήμα στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική με βάση τους στόχους που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελόνης το 2002 από την άποψη αυτή θα ήθελα να σας αναφέρω την πρόταση της οδηγίας για τη μητρότητα, ε, για την οποία θα επιληθεί ως ονόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνούμε με την, μια πρόταση που θα προστατεύει τη γυναίκα και τα δικαιώματα των ε, γυναικών που έχουν ε, γεννήσει, λεχώνων και γαλα, και γαλαχουσών μητέρων. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε το θέμα της διάρκεια της άδεια μητρότητα και της ε, ε, αμοιβή, την εξασφάλιση των εργατικών δικαιωμάτων των γυναικών ανάμεσα στην εγκυμοσύνη και στο τέλος της άδεια μητρότητας και φυσικά στην δυνατότητα επιλογής για τη στιγμή έναρξης της άδεια μητρότητας. Θα πρέπει επίση να γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα που ήταν 17,6% στην Ένωση το 2007 μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και αυτό το θέμα της μείωσης αυτού του μισθολογικού χάσματος είναι ένα ακόμη από τα θέματα που θα πρέπει να συμπεριλάβει με αποφασιστικότητα η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική. Γιατί θέλουμε όλο και περισσότερες γυναίκες να εργάζονται, αλλά όχι με χαμηλότερες αποδοχές από τους άντρες. Αντίθετα, θέλουμε να εδραιώσουμε ε, δεν θέλουμε να εδραιώσουμε ένα, μια νέα μορφή εκμετάλλευση που θα είναι αποδεκτή. Το μισθολογικό χάσμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μια αγορά εργασία που ε, μεταχειρίζεται με δυσμενή τρόπο τις γυναίκες. Γι' αυτό και θα πρέπει να εκφράσουμε τη δέσμευση και την αφοσίωση όλων των κρατών μελών προκειμένου να καταπολεμηθούν κάποια στερεότυπα των δύο φύλων και να αρθούν τα εμπόδια για την επαγγελματική ε, εκπλήρωση και των γυναικών και θα πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες σε επίπεδο διαπαιδαγώγησης. Η πλήρη ενσωμάτωση των γυναικών στον νέο μοντέλο απαιτεί μία συνυπευθυνότητα σε ό,τι αφορά την άσκηση της λήψη αποφάσεων στο πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα. Πέραν του κριτηρίου της δικαιοσύνης και του κριτήριου της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ε, συνηγορούν υπέρ της άποψης να δώσουμε και στις γυναίκες τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες για να έχουν πρόσβαση σε ηθήνουσες θέσεις πολιτικές και επιχειρηματικές. Γι' αυτό και θα πρέπει να προωθήσουμε την παρουσία των γυναικών σε ηγετικέ θέσεις των διοικητικών συμβουλίων και σε επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Κυρίε και κύριοι, η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σημαίνει κατά ανάγκη η προσπάθεια εκρίζωσης και της βίας μεταξύ των δύο φύλων. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί την πιο βάναυση εκδήλωση ε, μιας παιδείας και ενός πολιτισμού της ανισότητας και είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς έχει τις ρίζες τους όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι μια πραγματικότητα μπροστά στην οποία δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Με αυτόν τον τρόπο θα θέσουμε την καταπολέμηση τέτοιου είδους βίας στις πολιτικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου του 2002, των διαφόρων ψηφισμάτων που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1986 και με βάση το φύλλο πορείας για την ισότητα ανδρών και γυναικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, μπορώ ήδη να σας αναγγείλω ότι φροντίζουμε να καταρτήσουμε ένα σχέδιο συμπερασμάτων για την απάλληψη της βίας κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υποβάλουμε αυτό το σχέδιο στο επόμενο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Μαρτίου. Είναι ένα ευρύ σχέδιο συμπερασμάτων που καλύπτει όλους τους απαραίτητους παράγοντες για να καταργήσουμε, για να απαλείψουμε αυτή τη βία μεταξύ των δύο φύλων. Περιλαμβάνει κάποια σοφορονιστικά μέτρα και μέτρα προστασίας, αρρωγή στα θύματα, αλλά και πρόληψη και συνειδητοποίηση της κοινωνίας, αφύπνιση της κοινωνίας. Και όλα αυτά μέσω της κατάρτισης μιας κοινή στρατηγικής μεταξύ των 27 χωρών μελών. Γιατί αυτό είναι το κλειδί, μια και έχουμε ένα κοινό πρόβλημα και η λύση που θα επιλέξουμε θα πρέπει να στηρίζεται σε κοινά σημεία αναφοράς. Στο σχέδιο αυτό καλύπτουμε τα διάφορα είδη που υφίστανται οι γυναίκες εξαιτία του φίλου τους και της ε, βίας σε συναισθηματικό επίπεδο, του σωματοπορίου για σεξουαλική εκμετάλλευση, που είναι μια απαράδεκτη μορφή δουλείας που καταστρατηγεί τα θεμελιώδη δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει με μεγάλη αποφασιστικότητα να προσπαθήσουμε να την πατάξουμε. Θα ήθελα συνοπτικά να σας, περιλάβω, να σας απαριθμίσω κάποια μέτρα αυτού του σχεδίου συμπερασμάτων. Προτείνουμε για παράδειγμα την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη βία των φύλων. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την εφαρμογή κάποιων δικτών, τη συγκέντρωση στοιχείων με βάση μια κοινή μεθοδολογία την ανάλυση για την ε, δημιουργία γνώσης για τα χαρακτηριστικά της διάστασης της βίας κατά των γυναικών και για την ενημέρωση για τις καλύτερες πρακτικές ε, πάταξης αυτής της ε, βίας και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και πέραν των ορίων της. Και όλα αυτά σύμφωνα με το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου του 2009 σε σχέση με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης για το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά την ε, αρρωγή και προστασία στα θύματα της ε, βίας των φύλων, θα ήθελα να αναφέρω ότι στο πρόγραμμα δράσης του προγράμματος Στοκχόλμης βασιζόμαστε στην ε, υποστήριξη 12 χωρών μελών σε ό,τι αφορά την πρόταση οδηγίας Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Προστασίας. Έτσι, θα μπορούν οι γυναίκες που είναι θύματα βίας από τους συντρόφους που λαμβάνουν ε, ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που προσφέρει το κράτος το οποίο εξέδωσε αυτό το ένταλμα προστασίας. Θέλοντας να δώσουμε μια εναρμονισμένη λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις γυναίκες που είναι θύματα αυτών των εγκλημάτων, προτείνουμε στο σχέδιο συμπερασμάτων την ε, θέσπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ενιαία και δωρεάν Ευρωπαϊκής Γραμμής Κλήσης αρρωγής προς τα θύματα της βίας των φύλων. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε υποστήριξη για αυτή την πρωτοβουλία. Και όπως σας είπα, ήδη η Ευστρία, η Φιλανδία, η Σουηδία και η Πορτογαλία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και την υποστήριξή τους για την πρωτοβουλία αυτή. Το έτος 2010 ανακηρύσσεται ως το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και, της, και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα στραφούν οι στόχοι της Ισπανικής Προεδρίας. Για παράδειγμα, έχουμε την πρόταση οδηγίας για την ίση μεταχείριση που εξετάζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επεκτείνουμε και πέραν του εργατικού πλαισίου την προσπάθεια καταπολέμησης κάθε μορφής μεταχείρισης στα πλαίσια του άρθρου 19 του, της Νέας Συνθήκης της Λισαβόνας. Έτσι, λαμβάνουμε τη σκητάλη από τις προηγούμενες προεδρίες, τη Σουηδική και τη Γαλλική, και με βάση το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της Δευτέρας Απριλίου προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο προστασίας κατά της διακριτικής μεταχείρισης για λόγους φύλου, αναπηρίας, φιλετικής προέλευσης, εθνικής προέλευσης, γενετήσου προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκείας ή λατρείας. Βέβαια, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ε, πολλές επιφυλάξεις για το σχέδιο αυτό. Κατά τη γνώμη μας όμως είναι απαράδεκτο σε αυτή την κοινωνική Ευρώπη και Ευρώπη των δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζονται στη συνθήκη της Λισαβόνας και στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι αδιανόητο να δίνουμε διαφορετική λύση στη διακριτική μεταχείριση ανάλογα με την αιτία που την προκαλεί. Το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών γιατί συνεχίζονται. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου παρουσιάζοντας κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν στο εξάμεινο της Ισπανική Προεδρίας. Για παράδειγμα, θα διοργανωθεί το Ευρωπαϊκό Φόρουμ πεκίνος 15 στο Κάδι, 4 και 5 Φεβρουαρίου. Εκεί και οι κυβερνήσει των 27 χωρών μελών, τα κοινωτικά θεσμικά όργανα και η κοινωνία των πολιτών θα εγγύψουμε στις προτάσεις που έγιναν τα 15 χρόνια που πέρασαν από την πλατφόρμα δράση του Πεκίνου με βάση την έκθεση της Σουηδικής Προεδρίας. Το φόρμα αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε και την Πρόεδρο της Επιτροπής σας και τους ε, συντονιστές ε, και εκπροσώπους των κομμάτων. Στις 25 και 26 Μαρτίου θα γίνει στη Βαλένσια το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ισότητας. Εκεί θα ασχοληθούμε με τις πολιτικές ισότητες στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο που προσπαθούμε να ε, σχεδιάσουμε για την Ευρώπη. Επίσης θα έχουμε την πέμπτη σύνοδο ε, γυναικών από την Ισπανία και την Αφρική για ένα καλύτερο κόσμο. Εκεί θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το πρόγραμμά μας για την ισότητα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ προσβλέποντα σε μια επικοδομητική και καρποφόρα συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου τη Ισπανική Προεδρία. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση. Αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι εξαιρετικά εντατικές οι δραστηριότητες στον τομέα μας ε, επί Ισπανικής Προεδρίας και ευελπιστούμε σε μια αγαστή συνεργασία ε, ανάμεσα στην Προεδρία και την Επιτροπή μας. Υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοι που θα ήθελαν να υποβάλουν ερωτήματα. Ας ακούσουμε κάποιες από διάφορες πολιτικές ομάδες και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Η κυρία Μπάουερ θα πάρει πρώτη το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άπειρε ερωτήσει έχω υπόψη μου, αλλά θα περιοριστώ μόνο σε δύο για να επιτρέψω και στου λοιπού συναδέλφου να λάβουν το λόγο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ καταρχά για την ευκαιρία που μα προσφέρετε για ανταλλαγή απόψεων. Καλώ ήρθατε. Ελπίζω δε αυτή η συνάντηση να μην είναι ε, και η τελευταία μας. Θα ξαναπούμε σύντομα. Μιλήσατε νωρίτερα λοιπόν για τις ε, διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη διαφορετική μεταχειριστή. σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε να βελτιώσετε την συνειδητοποίηση, να ε, ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο. Εμείς είδαμε ότι υπάρχει μια πρόταση, μια ιδέα μάλλον για μια νέα πρόταση νόμου. Ή καλύτερα μια μελέτη για το πώς στην πράξη εφαρμόζεται η νομοθεσία. Το έχουμε δει αυτό ήδη στην πράξη. Ξέρουμε πολύ καλό ότι η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό. Άρα, ε, προφανώς, τα μέσα τα νομοθετικά δεν επαρκούν και θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά τους. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Ξέρω ότι μόνο νομοθεσία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Επίσης, αναφέρεται ότι θα πρέπει να ανανεωθεί η κοινωνική ατζέντα, το κοινωνικό μας πρόγραμμα. Πώς θα γίνει αυτό. Άλλη μια παρατήρηση, η ερώτηση. Μιλήσατε για το, ε, για την, για το Ευρωπαϊκό Διάταγμα προ... Ένταλμα Προστασίας. Πώς θα το προτείνετε, με τι μορφή ακριβώς, θα ξεκινήσετε από την πράσινη βίβλο, θα έχετε μια πρόταση πιο συγκεκριμένη, πιο άμεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Η κυρία Τόμψεν τώρα θα πάρει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Υπουργό για την διατύπωση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας της. Πρέπει να πω ότι για μας την Επιτροπή ε, δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών είναι πηγή ελπίδα στο ότι η ίση μεταχείριση αποτελεί προτεραιότητα για την Ισπανική Προεδρία. Πολλές ερωτήσεις λοιπόν δεν ήθελα και εγώ να διατυπώσω, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο θέμα της βίας βάρος των γυναικών. Η Ισπανία είναι από τα κράτη της Ευρώπης εκείνο με τα περισσότερες εμπειρίες ως προς την ε, υπόθεση αυτή. Έχει κάνει έρευνες πολλές, μελέτες, έχει η αστυνομία της ε, πολύ ε, πείραση λέξη. Ερώ λοιπόν πώς βλέπετε χάρη στην εμπειρία που διαθέτει η Ισπανία να επιλύεται ή να αντιμετωπίσετε μας περιπτώσει το πρόβλημα αυτό. Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε. Μπορεί να υπάρξει μια οδηγία ενδεχομένως για την αντιμετώπιση της βίας εις των γυναικών. Ευχαριστώ. Κυρία Χιμένας, παρακαλώ. Κυρία Χιμένες, ε, mm, Θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής των Γυναικών αλλά και προσωπικά να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην Επιτροπή μας. Από τότε που ανέλαβα το περασμένο Ιούλιο τα καθήκοντά μου, έθεσα ως προτεραιότητά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προσπάθεια αναχέτησης της βίας κατά των γυναικών. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να λάβει κάποια μέτρα για να προστατεύσει τα θύματα. Γι' αυτό στις 19 Οκτωβρίου εγκρίθηκε ένα σχέδιο ψηφίσματος για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ό,τι αφορά το χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Και μάλιστα τότε ζήτησε από την Ισπανική Προεδρία να προωθήσει την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό ένταλμα προστασίας των θυμάτων της βίας στο φύλου, για να επεκταθούν και πέραν της εθνικής επικράτειας τα μέτρα αυτά. Οι τροπολογίε μου τελικά εγκρίθηκαν και συμπεριλήθηκαν στο τελικό ψήφισμα για το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. και θα ήθελα να συγχαρώ την Ισπανική Προεδρία γιατί πρόθεσε το σχέδιο αυτό για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα προστασία και το θεώρησε και προτεραιότητα. Τι μηχανισμού θα προτείνει η Ισπανική Προεδρία ώστε αυτό το Ευρωπαϊκό Ένταλμα να προστατεύει και αποτελεσματικά τα θύματα τη βιότητα. Πιστεύετε ότι στη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, ε, δράτω με τις ευκαιρίες για να σας ρωτήσω τη γνώμη της Ισπανικής Προεδρίας και το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη δυσανάλογη έξαρση της γυναικείας ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στην ε, δική μου γενέτερα, την Ανταλουσία που είναι και δική σας, ε, η γυναική ανεργία φτάνει στο 27% και οι γυναίκες υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες του να πρέπει να αναλαμβάνουν τα οικογενειακά βάρη ενώ όλα τα μέλη της οικογένειας ε, είναι άνεργα. Η Ισπανική Προεδρία σκοπεύει να υιοθετήσει κάποια μέτρα για να προστατεύσει τις έγκυες γυναίκες που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης χάνουν τις δουλειές τους και αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον προσπαθώντας να συνδυάσουν τον επαγγελματικό και τον οικογενειακό τους βίο. Θα προωθήσετε κάποιες ενισχύσεις προς τις οργανώσεις και τις ενώσεις που δίνουν μάχη για να βοηθήσουν τις γυναίκες που θέλουν να τεκνοποιήσουν αλλά που πολλές, σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται μόνες τους και αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μποσκούτ τώρα. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση ως προς την οδηγία για την ισότητα μεταχείρισης. Με χαρά βλέπω ότι κρίνεται το θέμα αυτό επίσης της προτεραιότητας και εσείς ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε τη Σύνοδο Κορυφή για την ισότητα ευκαιριών ε, στην ε, Σουηδία πριν από ένα-δύο μήνε. Ε, και από τι ερωτήσει που έχω να σας υποβάλω κάταρχα, θα ήθελα να μας πείτε για τη Σύνοδο Κορυφή αυτήν της ισότητας φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση η Βελγική Προεδρία να κλείσει το θέμα αυτό αλλά από την άλλη μας λέτε εσείς ότι στο τέλος της Τρόικα μόνο θα είναι όριμο προς ε, ολοκλήρωση το ζήτημα αυτής της οδηγίας. Γιατί να καθυστερήσουμε τόσο και τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να λάβει η Ισπανική Προεδρία έτσι ώστε να καταλήξει σε μια ισότητα μεταχείρισης. Αυτό που επίσης θα ήθελα να μάθω. Και παρακαλώ μου δώστε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πριν από, ένα, πριν από χρόνο πάλι τα ίδια θέματα συζητήσαμε, τις μεγάλες ε, ε, προκλήσεις της θρησκείας, της σεξουαλικής, ε, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή επιλογών του, των αναπηριών. Τα τέσσερα μεγάλα θέματα που απασχολούν τις ειδικέ ομάδες πληθυσμού και τις γυναίκες ιδιαίτερως και ε, εδώ είδαμε ότι δεν υπάρχει επαρκής παροχή υπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε να αναλυφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Η Ισπανική Προεδρία τι σκοπεύει να κάνει. Θα προχωρήσει ή θα πρέπει πάλι να περιμένουμε μέχρι και την Ουγγρική Προεδρία. Έχουμε καθυστερήσει πολύ εδώ μεταξύ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Εστρέλα, η αντιπρόεδρός μας τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για την παρουσίαση που κάνατε με όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά επίσης να ε, συγχαρώ την ε, Ισπανική Προεδρία διότι έχει αναδείξει σε προτεραιότητα αυτά τα θέματα της ισότητας των δύο φύλων και κυρίως αυτή την δημιουργία του παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ε, έχω το ρόλο της εισηγήτριας για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητος και παρότι θα είχα και άλλες ερωτήσεις να σας υποβάλω, θα επικεντρώσω την προσοχή μου σε αυτό το θέμα, διότι είναι αυτό που με αφορά μεσότερα από όλα τα υπόλοιπα και εξάλλου και εξαιρετικά επίκαιρο αυτό το θέμα, διότι ε, σήμερα θα συζητήσουμε μάλιστα τις τροπολογίες ε, που υπευλήθησαν ε, από διάφορους, από διάφορους βουλευτίνες. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Ισπανική Προεδρία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην λόγω οδηγία όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο της, που έχει σημασία για την προστασία των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και επειδή αναβαθμίζει τον ενδυνάμει ρόλο των γυναικών κατά την έξοδο από την οικονομική κρίση. Και μιλήσατε για συνυπευθυνότητα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο μιας ε, ρηξικέλευθης ε, πρότασης ε, του, της έκθεσης, δηλαδή ομιλώ για την άδεια πατρότητας. Δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπεται μόνο άδεια μητρότητας. Και υπάρχει και μία άλλη οδηγία για την γονική άδεια. Και παρότι στην πλειοψηφία των κρατών μελών, με εξαίρεση την Ιταλία και τη Γερμανία, προβλέπεται στην οικία νομοθεσία η άδεια πατρότητας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υφίσταται πρόβλεψη. Να λοιπόν η χρυσή ευκαιρία για να καλύψουμε αυτό το κενό και για να εξυγχρονίσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε με αυτή τη μορφή να προάγουμε και την συμφιλίωση ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή και προσωπική ζωή. Αυτό θα το επιτύχουμε μόνο με τον σωστό κατημερισμό των ευθυνών στο ιστορικό κάθε οικογένειας. Η Ισπανική Προεδρία στο Συμβούλιο θα υπεραμεινθεί αυτή τη θέση, δηλαδή να συμπεριληφθεί μέσα στην εν λόγω οδηγία και η μέρημνα για την άδεια πατρότητα. Σα ευχαριστούμε και πάλι συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία για την Προεδρία σα. Ευχαριστούμε κυρία Εστρέλα. Ο κύριος Δρομέβα τώρα και κατόπιν θα ακούσουμε την Υπουργό για να απαντήσει στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Ο κύριος Ρομίβας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά και να σας επενέσω για την σημασία που έχει και το συμβολισμό που έχει παρουσίαση. γιατί σπάνια έχουμε υπουργούς που έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα και προτεραιότητα αυτά τα θέματα. Γιατί πολλέ φορέ είχαμε υπουργού που είχαν ε, στα καθήκοντά του και αυτό το θέμα τη ισότητα, αλλά ως και προτεραιότητα πρώτη φορά, πρώτη φορά το βλέπουμε και σα συγχαίρουμε θερμά. Είναι υπερφορτωμένο το πρόγραμμα τη ισπανική προεδρία. Θα ήθελα να πω και εγώ ότι, όπω είπε η κυρία Στρέλε, είμαστε υπέρ της άδεια πατρότητα. Και όχι μόνο είμαστε υπέρ τη ανάγκη της άδεια πατρότητας, αλλά της υποχρέωσης που έχουν οι άνδρες να αναλαμβάνουν και αυτή το ρόλο της ανατροφής των παιδιών. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η άδεια πατρότητας θα πρέπει να κατοχυρωθεί και να συμπεριληφθεί στην οδηγία για την άδεια μητρότητας. Αλλιώς ε, θα προσθεθεί μία ακόμη διακριτική μεταχείριση κατά των ε, γυναικών. Και θα πρέπει να είναι ε, μία εναλλακτική πρόταση για την άδεια μητρότητας και συμπληρωματική. Και Σα διαβεβαιώ κύριε Υπουργέ ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ η υπέρμαχη αυτή τη θέση για την άδεια πατρότητα. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τι πολλαπλέ μορφέ μεταχείριση. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει προσκρούσει ένα διέξοδο στο Συμβούλιο, γιατί κάποιε χώρε αντιμετωπίζουν δυσκολίε με την οδηγία αυτή. Μπορείτε να μας πείτε σε τι φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, ποιες είναι οι συγκεκριμένες δυσκολίες και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Αν δικαιολογείται δηλαδή κάποια αισιοδοξία ότι αυτό το θέμα θα διεκπαιρεωθεί στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Ή τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς θα μπορούσε να συμβάλλει για να ξεφύγουμε από αυτήν την αποτελμάτωση στην οποία έχει κολλήσει η οδηγία αυτή. Τέλος. Στο πλαίσιο της κρίσης ε, είναι προφανές ότι έχουμε πολλά μέτρα με στόχο την ανάκαμψη της οικονομίας με συγκεκριμένα προγράμματα δράσης. Αυτό που λείπει πολλές φορές είναι η προοπτική των δύο φύλων στα μέτρα αυτά. Γιατί πολλούς από τους τομείς που κανονικά θα πρέπει να είναι τομείς ε, εχμής και θα πρέπει να είναι το λάβαρο και το προπύργιο αυτής της οικονομικής ανάπτυξης είναι τομείς που κατά παράδοση δεν χαρακτηρίζονται από σημαντική συμμετοχή και παρουσία των γυναικών. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, η υποστήριξη δηλαδή των γυναικών για να γίνουν πιο αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα για την ανάκαμψη και την έξοδο από την κρίση. Τώρα, το θέμα της εξατομίκευσης των ε, συντάξεων. Σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι συντάξεις εξαρτώνται από, την, από το χαρακτηρισμό σύζυγος του. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και επίγει να το ρυθμίσουμε το συντομότερο δυνατό. Το θέμα της εξατομίκευσης των συντάξεων είναι θέμα όχι μόνο πολιτικό αλλά κυρίως κοινωνικό. Και ένα θέμα διεθνούς πολιτικής. Έχουμε μια προεδρία που θα πρωτοστατήσει σε συμφωνίες με τη Λατινική Αμερική, θα διοργανώσει πολλές διασκέψεις κορυφής με, στη Μεσόγειο, με τις ασιατικές χώρες και στις συμφωνίες σύνδεσης υπάρχουν μελέτες επιπτώσεων, οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών. Σε μια πρόσφατη έκθεση προτάθηκε η μελέτη επιπτώσεων και υπό το πρίσμα των δύο φύλων. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι ε, δέχτηκε μάλλον ικανοποιητικά αυτή την πρόταση. Ερωτώ λοιπόν, στι συμφωνίε σύνδεση που διαπραγματεύεστε, είναι δυνατόν ή απαραίτητο να προβληθεί και από το θέμα της επίπτωσης που έχουν οι συμφωνίες αυτές στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Στην Κεντρική Αμερική, για παράδειγμα, στη Λατινική Αμερική, στη Μεσόγειο, είναι σημαντικό αυτό το θέμα της ισότητας των φύλων. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα μπορούσε να περιληφθεί και αυτή η απαραιτητο να προβληθει και απο το θεμα της επίπτωση που εχουν οι συμφωνιες αυτες στο θεμα της ισοτητα των δυο φυλων στην κεντρικη αμερικη για παραδειγμα στη λατινικη αμερικη στη μεσογειο ειναι σημαντικο αυτο το θεμα της ισοτητα των φυλων πιστευετε λοιπον οτι θα μπορουσε να περιληφθει και αυτη η διασταση στι συμφωνίε σύνδεση γιατί πολλές φορές και αθέλητα τους μάλιστα οι συμφωνίες είδησης δημιουργούν δυσμενείς επιπτώσει για την ισότητα των φύλων. Ευχαριστούμε κύριε Ρωμέβα. Θα δώσουμε το λόγο στην Υπουργό για να απαντήσει στον πρώτο γύρο ερωτημάτων. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής μας για τις παρατηρήσεις τους. Θα προσπαθήσω να ομοδοποιήσω κάπως τις απαντήσεις. Αναφέρθηκε το μισθολογικό χάσμα. Χαίρομαι που διαπιστώνω το ζωηρό ενδιαφέρον που δείχνει η Επιτροπή σας για την μείωση αυτού του μισθολογικού χάσματος, γιατί το μισθολογικό αυτό χάσμα αποτελεί μια απαράδεκτη μορφή διακριτικής μεταχείρισης βάρος των γυναικών. Και όλες μας οι προσπάθειες είναι λίγες. Θα πρέπει να τις εντείνουμε και να εντείνουμε και τη συνεργασία μας προκειμένου να γεφυρωθεί αυτό το άδικο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και δύο εδώ είναι οι παράγοντες κλειδιά. Το γεγονός ότι θα έχουμε κάποιους ελεκτικούς μηχανισμούς για να αποφύγουμε καταστρατήγηση της ισχύωσης νομοθεσίας που απαγορεύει την ύπαρξη τέτοιων μισθολογικών διαφορών. Για παράδειγμα, για να σας δώσω το συγκεκριμένο παράδειγμα της ε, πατρίδας μου, της Ισπανίας. Έχουμε συνάψει μια συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Απασχόλησης και Υπουργείου Ισότητας σε ό,τι αφορά την εξακρίβωση των μισθολογικών διαφορών στις διάφορες επιχειρήσεις. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κάποια φαλοκρατικά στερεότυπα στην παιδεία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τώρα, τι συγκεκριμένα θα πράξει η Ισπανική Προεδρία στον τομέα αυτό. Αυτή ήταν η συγκεκριμένη ερώτηση της κυρίας Μπάουερ. Θα προσπαθήσουμε στην στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών ε, Ισότητας που θα γίνει στις 25 και 26 Μαρτίου στη Βαλένθια θα υποβάλουμε την προκαταρκτική έκθεση για τις μισθολογικές διαφορές που θα αποτελέσει και τη βάση για την Βελγική Προεδρία που θα αναγάγει αυτό το θέμα της καταπολέμησης των μισθολογικών διαφορών σε ύψιστη προτεραιότητα το αγώνα τη για την αποκατάσταση τη ισότητα των ευκαιριών. Και αυτό το στόχο έχει και το τρίο, η συνεργασία μεταξύ των τριών προεδριών, για να εξασφαλίσουμε μια συνέχεια και μια καλύτερη εφαρμογή των ε, κοινών μα προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασία. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται το στόχο της Ισπανικής Προεδρίας ώστε η βία των φύλων αποτελέσει πρωταρχική προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας και ελπίζουμε να εξασφαλιστεί συνέχεια και από την επόμενη Προεδρία. Και σίγουρα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασία είναι πρωταρχικό μα στόχο, γιατί επεκτείνουμε έτσι την προστασία των γυναικών που είναι θύματα τη βία ε, και να αναγνωριστούν κάποια ε, μέτρα δικαστικά που λαμβάνονται στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία, ώστε να μην επιτρέπεται ατιμορρησία των ε, αυτούργων της βίας. Ε, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Το γεγονός ότι υπάρχει ένταλμα απομάκρυση από το θύμα ε, θα πρέπει να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και ελπίζω ότι εκ περιτροπής Προεδρία με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση αυτή οδηγία, που θα αποτελέσει σημαντική πρόοδο ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό χώρο ασφάλεια, ελευθερία και δικαιοσύνη και τη καταπολέμηση ε, τη βία, να ευοδοθεί. Γιατί και το Συμβουλίο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ε, ασχολείται με το θέμα αυτό σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνη και το Υπουργείο Ισότητα Ευκαιριών. Έχουμε στενή συνεργασία για τα θέματα αυτά, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Προστασία, γιατί είναι πολύ σημαντικό στην προστασία αυτή να συμπεριληφθούν όχι μόνο θύματα άλλων εγκλημάτων, αλλά και θύματα τη βία ε, στο σπίτι των φίλων. Τώρα, ποια ήταν η Ισπανική Προεδρία σε θέματα καταπολέμησης ε, της βίας κατά των γυναικών. Στην Ισπανία είχαμε ένα σημαντικό σημείο καμπής με την ε, έγκριση του Γενικού Νόμου κατά της βίας των φύλων. Έτσι εξασφαλίστηκε μεγαλύτερη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των πολιτών και υπήρξε σημαντική συνένεση γιατί ο νόμος αυτός εγκρίθηκε ομόφωνα στην Ισπανική Βουλή και πρόσφατα η Επιτροπή Ισότητας ε, της Βουλής των Αντιπροσώπων της ε, Ισπανίας τάχθηκε υπέρ του γενικού αυτού νόμου στη συνδιάσκεψη των Προέδρων των Αυτονομιών και εκεί υπήρξε συνένεση για την πάταξη της βίας των φύλων και νομίζω ότι αυτός ο συντονισμός, αυτή η σύμπνη, αυτή η ομόνια, η συνεργασία και αυτό το κοινό πνεύμα έχει κάποιο αποτέλεσμα και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ξεριζώσουμε αυτή την κοινωνική μάστιγα που είναι η βία στα, μεταξύ των δύο φύλων. Πάντως ε, η συμμετοχή των πολιτών ήταν ε, το σημείο καμπής σε αυτή την πορεία. Καταφέραμε να εξαγάγουμε το θέμα από τον ιδιωτικό χώρο στο δημόσιο χώρο. Το θέμα πια δεν είναι το θέμα τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι, τι συμβαίνει μέσα στο ζευγάρι, τι συμβαίνει στα εσωτερικά του κάθε οίκου είναι θέμα κοινωνικό. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, γιατί όλοι φέρουμε ευθύνη για την πάταξη αυτού του προβλήματος. Στην Ισπανική κοινωνία υπήρξε σημαντική πρόοδος και στο θέμα της πρόληψης και στο θέμα της διαπαιδαγώγησης. Όλο και περισσότεροι νέοι ευαισθητοποιούνται σε θέματα πολίτη και αγωγής του πολίτη και προστασίας και καταπολέμησης της βίας και μάλιστα ε, είχαμε, θέσαμε 3.000 ε, συσκευές εντοπισμού ε, της απόστασης στα δικαστήρια της Ισπανίας για την προστασία των θυμάτων. Επίσης θέλουμε να έχουμε ομοιόμορφες και ομοιογενείς πληροφορίες για όλα τα εγκλήματα. Έχουμε διάφορες πτυχές υγειονομική, αστυνομική, δικαστική. Δεν θέλουμε οι γυναίκες, ε, εκτός από τον πόνο που έχουν ε, και την κατάσταση του θύματος, να πρέπει να αντιμετωπίζουν και μια φόρητη γραφειοκρατία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις αποκλειστικέ αποκλειστικά δικαστήρια και για το θέμα αυτό και 1.500 ε, αστυνομικές, αστυνομικούς που ασχολούνται με το θέμα αυτό, 3.000 γυναίκες που απασχολούνται στην ε, τηλεαρρωγή πάνω από 20.000 γυναίκες ε, δέχονται αυτό το ενεργό επίδομα ένταξης, πολύ σημαντικό για να εξασφαλιστεί ένα είδος οικονομικής ανεξαρτησίας. Έχουμε το τηλέφωνο 016 που είναι η δωρεάν γραμμή που έχουν τα θύματα στη διάθεσή τους. Κάθε, καθημερινά λαμβάνουμε 200 κλήσεις σε αυτή τη γραμμή και μάλιστα έχουμε πάνω από 70.000 ε, φυλακισμένους που εκτίουν ποινές εξαιτία διάπραξη τέτοιου εγκλήματος και νομίζω ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος στο δρόμο της εκρίζωσης αυτής της μάστιγας και σε καμία περίπτωση θα πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί ούτε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας θα πρέπει με εντυμότητα και πυγμή να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πάντω το 2009 μπορούμε να πούμε ότι 55 γυναίκες ε, έχασαν τη ζωή του από τη φαλοκρατική βία. Ε, βέβαια είχαμε 21 γυναίκε λιγότερε από το 2008. Παρ' όλα αυτά τα θύματα εξακολουθούν είναι πολλά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα. Έχουμε 55 επιπλέον λόγου να συνεχίσουμε την προσπάθειά μα και το έργο μα στο τομέα αυτό. Αλλά έχουμε και 21 λόγου που μα δημιουργούν ε, ελπίδα και αισιοδοξία. Και με την αρρωγή ε, της κοινωνίας ε, των πολιτών και με τη συνένεση που διαμορφώθηκε μεταξύ των πολιτικών ε, δυνάμεων και με καλό συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων πιστεύω ότι μπορούμε να θέσουμε τέρμα στη βία μεταξύ των φύλων. Αλλά φυσικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πιο ισότιμη κοινωνία, να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στη διαπαιδαγώγηση, στην αφύπνιση, στη συνειδητοποίηση και να έχουμε μια συνολική προοπτική. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος μας. Μια ολιστική πρόπτικη αυτού του προβλήματος. Σε ό,τι αφορά τώρα την οδηγία, στόχο έχουμε να υποβάλουμε το σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Μαρτίου, της 8ης και 9ης Μαρτίου. Τα συμπεράσματα αυτά θα συμπεριλαμβάνουν και το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών με αυτή τη συνολική προοπτική. Στα συμπεράσματα αυτά γίνεται λόγος για πρόληψη, γίνεται λόγος για προστασία, για απομάκρυνση των αυτούργων, για την τιμωρία των αυτούργων, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Επίσης έχουμε την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας, την ενιαία Ευρωπαϊκή Γραμμή Δωρεάν Κλήσης για τα θύματα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά βήματα, αποφασιστικά βήματα και ελπίζω να εγκριθεί αυτό το σχέδιο συμπερασμάτων και έχουμε στενή συνεργασία για το θέμα αυτό με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί το Συμβούλιο μόνο μετά από πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να λάβει κάποιες νομοθετικέ αποφάσεις. Έχουμε λοιπόν επίγνωση ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εγκύπτει στο θέμα εκπονώντας μία έκθεση για την εναρμόνιση των διαφόρων νομοθεσιών. Ελπίζουμε από την έκθεση αυτή να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στις εθνικές νομοθεσίες και να σημειώσουμε πρόοδο. Πάντως η Ισπανία είναι προσιλωμένη σε αυτό το στόχο και ε, έχει τη βία, την πάταξη της βίας ε, μεταξύ των φίλων στο επίκεντρο της Προεδρίας και ως ύψιστη προτεραιότητά της. Θέλουμε αυτό το θέμα να το προαγάγουμε και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκαν και κάποιες παρατηρήσεις για την γυναική ανεργία, για το υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών. Σε μια πρώτη φάση η κρίση έπληξε περισσότερο την ε, ανεργία στους άνδρες. Τώρα τελευταία όμως είχαμε παρόμοιες ανησυχητικές τάσεις και στις γυναίκες. Στην Ισπανία είχαμε 25,4% ανεργία μεταξύ το Δεκεμβρίου 2008 και Δεκεμβρίου 2009 και στο επίπεδο των γυναικών ήταν 23,9%. Δηλαδή είχαμε μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Στους άνδρες είχαμε 27,6%, στις γυναίκες 23,9%. Πάντως, ο σχεδιασμός αυτής της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Θα πρέπει επίσης να μειωθούν οι μισθολογικές διαφορές. Θα πρέπει με αποφασιστικό τρόπο να προωθήσουμε την συνυπευθυνότητα. Να έχουμε κοινού ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει να συμφιλιώσουμε καλύτερα τον επαγγελματικό και οικογενειακό βίο, να γίνει ένας καλύτερος και πιο ισότιμος καταμερισμός των οικογενειακών βαρών και της ανατροφής των παιδιών. Όλοι αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να περιληφθούν στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020, κάτι που αποτελεί βασικό σκοπό της Ισπανικής Προεδρίας. Ό,τι αφορά τις εγγύους και τα συγκεκριμένα μέτρα αρρωγής προς τις εγγύους. Θα ήθελα να πω ότι σίγουρα θα πρέπει να βοηθήσουμε τις εγγύους ε, για να συμπεριληφθούν στην αγορά εργασίας και να μπορέσουν ε, να συνδυάσουν με αρμονικό τρόπο την ε, οικογενειακή με την επαγγελματική του ζωή. Θα σας δώσω και πάλι το παράδειγμα της Ισπανίας. Το 2007 υιοθετήσαμε το νόμο για την ισότητα ανδρών και γυναικών που είναι το καλύτερο σχέδιο συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Και σήμερα οι έγκυες στην, γυναίκες στην Ισπανία τη χάνουν της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας κατά της απόλυσης. Έγινε κάποια βήματα για να αναγνωριστούν και οι περίοδοι ε, άδειας μητρότητας ως κανονικές περίοδοι εργασίας και εισφοράς, κοινωνικής εισφοράς. Και, και έγιναν κάποια, κάποιες τροποποίησεις στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Επίσης, ε, ε, έχουμε προτείνει το σχέδιο ΕΝΤΟΥΚΑ 0-3 προκειμένου να ε, αναλυθούν κάποιες φροντίδες ε, και να βελτιωθούν οι βρεφονιβιακοί σταθμοί για την φροντίδα των παιδιών από 0 3 χρόνια. Έχουμε το, την άδεια πατρότητας που είναι ανεξάρτητο από την άδεια μετρότητας και μάλιστα 80% των ε, ανδρών που γίνονται πατέρες εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα της άδειας πατρότητας. Δώσαμε έμφαση λοιπόν στη συνυπευθυνότητα, στον καταμερισμό των ευθυνών και στην ε, συμφιλίωση οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Νομίζω ότι έτσι βελτιώσαμε κατά πολύ τη θέση των εγγύων γυναικών στην Ισπανία. Σε ό,τι αφορά την ισότητα τη μεταχείριση και τη σχετική οδηγία για την ίση μεταχείριση, όπω σα είπα για την Ισπανική Προεδρία, αυτό ο στόχο θα είναι επίση κέριο και συνεργαζόμαστε με το τρίο την Ουγγαρία και το Βέλγιο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες δυσκολίες γιατί ορισμένες χώρες έχουν σοβαρές επιφυλάξεις, ορισμένες για την νομική βάση, γιατί προηγούμενα έχουμε. Δεν πρόκειται για κάτι καινοτόμο και άνευ προηγουμένου. Δεν είναι ότι με μια οδηγία θα, ξεπεράσουμε στο εργατικό επίπεδο το θέμα της ισότητας των ευκαιριών της ίσης μεταχείρισης. Είχαμε παρόμοιες οδηγίες, οπότε υπάρχει απόλυτα σωστή και κατάλληλη νομική βάση. Ούτε θέλουμε να σφετεριστούμε τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα θέματα κοινωνικής ασφάλειας, προστασίας, υγειονομικής περίθαλψης, παιδείας ή στέγασης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης ε, σε διάφορες υπηρεσίες θα πρέπει κανένας πολίτης, ε, ούτε άνδρας ούτε γυναίκα, να μην τη χάνει άνηση μεταχείρισης για οποιαδήποτε οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται. Επίσης, δεν θα πρέπει να είναι διαφορετική η μεταχείριση ανάλογα με την αιτία της ε, διαφοράς. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το λίκνο ορισμένων αξιών και δικαιωμάτων και αρχών. Βέβαια, πρόκειται για μια οδηγία. Δεν θα πρέπει να αρκεστούμε στο μη χείρον βέλτιστον προσπαθούμε να επιτύχουμε κάποια εναρμόνιση στο θέσιο, να προλιάνουμε κάποιο, κάπως το έδαφος, γιατί θα είναι πολύ απογοητευτικό να μην καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας έναντι οποιασδήποτε μορφής ε, άδικης ή άνης μεταχείρισης, γιατί η ίδια συνθήκη κατοχυρώνει την ίση μεταχείριση. Είναι γνωστέ οι δυσκολίε, αλλά δεν πρόκειται να παρατηθούμε, ούτε να συνθηκολογήσουμε. Δεν μπορώ φυσικά να προεξοφλήσω την έκβαση των διαπραγματεύσεων, πάντω ευελπιστώ ότι θα εξασφαλίσουμε και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη συνενοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πρόγραμμα αυτό και ελπίζω ο καθένας στην πατρίδα του να προωθήσει αυτό το θέμα και να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση και στην κατανίκηση των αντιστάσεων που παρουσιάζουν μερικές φορές ορισμένες χώρες μέλη. Σας ευχαριστούμε. για να το γνωρίζετε. Έχουμε άλλους εννέα συναδέλφους που θέλουν ε, να μιλήσουν. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Προσπαθήστε. Η κυρία Κλάς πρώτη και η κυρία Γκασίγια Πέρες στη συνέχεια. Κυρία Κλάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου. Μας ε, παραθέσατε μια σειρά πυροτεχνημάτων σε προτεραιότητες ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είναι καινούριο θέμα βέβαια και δεν βλέπω πουθενά καινούρια νέα μέτρα. Πώς δηλαδή σκοπεύει η Ισπανία συγκεκριμένα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Η Σέλφος Εστέλα ήδη ρώτησε τι γίνεται με την οδηγία για την προστασία της μητρότητας. Και τώρα και στη δεύτερη σας ε, απάντηση, στη δευτερολογία σας, μιλήσατε ακροθυγώς για την αγορά εργασίας. Εγώ βλέπω πολύ στενή σχέση μεταξύ της οδηγίας για την προστασία της μητρότητα και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που με τον οποίο θα χειριστούμε την ε, οδηγία. Η προστασία της μητρότητα σημαίνει προστασία της υγείας της μητέρας και επαρκή χρόνο για τους γονείς. Αλλά δεν θα ήθελα να αναμειχθούν τα θέματα υγείας της ε, μητέρας και της ε, άδεια μητρότητα που δεν είναι βέβαια 20 εβδομάδες και του χρόνου της γονικής άδεια. Η δε πρόσβαση στην αγορά εργασίας σημαίνει εμπλοκή και της οικονομίας και των επιχειρήσεων, αυτών που διαχειρίζονται τις θέσεις εργασίας. Πώς θα μπορέσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή και των ε, εργοδοτών. Επίσης, στις τοποθετήσεις σας μιλήσατε και για τη βία εις βάρος των γυναικών. Το παρατηρητήριο θα πρέπει κατά την άποψή μου να συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη και θα πρέπει και εμείς να παρακολουθήσουμε από πλευρά μας ε, την υπόθεση αυτή για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αλλά και για να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Και λίγο πριν από την παγκόσμια διάσκεψη για τη γυναίκα της Νέας Υόρκης, εκείνος είναι πέντε έτη, Κυρία Πρόεδρε, έχετε κάποια προτεραιότητα να πάρετε μαζί σας, να βάλετε μαζί στη βαλίτσα σας στη Νέα Υόρκη. Όχι όλες τις προτεραιότητες, μία ή δύο σοβαρές που να εκφράζουν τις Ευρωπαίες. Ίσως θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με τις γυναίκες σε περιοχές κρίσης επιπλέον και ίσως θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερως οι γυναίκες στην IT. Ευχαριστούμε. κυρία Κασία Πέρες τώρα και πριν πάρετε το λόγο, ήθελα να σα ενημερώσω ότι η προσκεκλημένη μα ε, θα πρέπει να φύγει σε 25 λεπτά στι 4.30. Αφήστε τη και λίγο χρόνο παρακαλώ για να μπορέσει να απαντήσει. Η κυρία Πέρες. Ευχαριστώ. Θα είμαι λακωνική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό μας για την παρουσία της στην Επιτροπή μας γιατί για μας είναι σημαντική αυτή η παρουσία. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω και για το πρόγραμμα που μας παρουσίασε. Γιατί όποιος δεν είναι φιλόδοξος στο έργο του, όποιος πιστεύει ότι ε, δεν έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει σε θέματα ισότητας, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που λέει το 52% του ευρωπαϊκού πληθυσμού είναι γυναίκες ε, και υφίστανται σοβαρές ε, περιπτώσεις άνηση μεταχείρισης, ιδιαίτερα στο τομέα της εργασίας μία παρατήρηση για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της βίας κατά των φύλων. Μας δώσετε πολύ σημαντικά στοιχεία για την Ισπανία για τη βία μεταξύ των φύλων. Χρειαζόμαστε και μηχανισμούς αλλά και γενικά στοιχεία από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επεξεργαστούμε κάποια κοινά εργαλεία και να πατάξουμε τη βία μεταξύ των φύλων. Στην πρότασή σας για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο προβλέπετε η συγκρότηση κάποιων κοινών μηχανισμών και εργαλείων για να ε, λάβουν σάρκα και οστά οι ευρωπαϊκές πολιτικές καταπολέμησης της βίας. Ευχαριστούμε κύριο Σταραμπέλα. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Υπουργέ. Μέχρι την ώρα που ήρθατε εδώ στην ε, αίθουσα νόμιζα ότι η ωραία του Κάδηξ είναι απλώς ένα πρόσωπο από την οπεράτα του Λόπες. Δεν ήξερα ότι υπάρχει στην πραγματικότητα τέτοια ομορφιά και να που τη βλέπω μπροστά μου. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που σα βλέπω εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε συγκεκριμένα προβλήματα όπω τη βία κατά των γυναικών, το, το pick-up ε, και άλλα. Ευχαριστώ ταυτόχρονα και την Ισπανική κυβέρνηση για τι προσπάθειε τη προσπάθειε για αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Και βεβαίως να σημειώσω ότι η Προεδρία σα με τις ψηλές προτεραιότητε που δίνει με των γυναικών έρχεται ε, την κατάλληλη στιγμή. Εγώ λοιπόν με την έκθεση που έχω προτείνω και την ε, θέσπιση έτους για την ε, αντιμετώπιση της βίας, κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές προσπάθησε να ορίσει τέτοιο ευρωπαϊκό έτος, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το θεώρησε σκόπιμο. Μείναμε λοιπόν χωρίς απάντηση, χωρίς ανταπόκριση στην υπόθεση αυτή και θα σας ρωτούσα εάν θα συμφωνούσατε μέσα στο πρόγραμμά σα να συμφωνήσετε με την θέσπιση ενό τέτοιου το φετινό είναι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με θέσπιση έτου ευρωπαϊκού δεν αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον ευαισθητοποιούμε τον κόσμο και ξεκινούμε την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σε ευχαριστώ πολύ με την ελπίδα ότι θα υποστηρίξετε την πρωτοβουλία αυτή. Ευχαριστούμε η κυρία Έρνστ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, μάλλον θα είναι Ανιαρή εποδός να πω ότι εδώ η Επιτροπή των Γυναικών χαίρει που σας βλέπει και χαίρομαι για τις προτεραιότητες και τη στράτευσή σας για τα θέματα των γυναικών. Πριν όμως έχουμε αρκετά προβλήματα ακόμα για να προχωρήσω. Έχουμε ζητήματα ως προς την ανισότητα, την μη τήρηση της αρχής δηλαδή, της ισότητας. Έχουμε να κάνουμε με αποφάσεις οι οποίες ε, ε, δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να αναλάβουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Έχουμε να κάνουμε επίσης με θέσεις, προτάσεις ε, ή πρακτικέ οι οποίε χωρί να είναι υποχρεωτικέ, δηλαδή χωρί να φέρουν τη γυναίκα σε μια κατάσταση υποχρεωτική, την αναγκάζουν ουσιαστικά να πάρει μια απόφαση που τη επιβάλλεται όμω και που είναι ει βάρο τη, ει τη ισότητα. Ερωτώ λοιπόν. Για τα κράτη-μέλη, συγκεκριμένα προγράμματα, ιδέες, μέτρα, για κυρώσεις ενδεχομένως όταν δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία, όταν δεν επιβάλλουν στις επιχειρήσεις τους ε, την νομοθεσία ή δεν επιβάλλουν τις κυρώσεις που θα έπρεπε να επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρης αρχές της ίσης ε, μεταχείρισης των εργαζομένων. Επίσης, ως προς την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και ε, κυρίως στις ε, ηγετικέ θέσει στι οποίε αναφερθήκατε, στα διοικητικά όργανα στα οποία αναφερθήκατε, όταν έχουμε τέτοια προβλήματα, Έχετε κάποιες ιδέες συγκεκριμένε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ένα διοικητικό συμβούλιο πορτίζεται σχεδόν αποκλειστικά από άντρε ή αποκλειστικά από άντρε, δεν είναι αυτοί διατεθειμένοι να ε, εκχωρήσουν μέρο τη εξουσία του. Τι συγκεκριμένα έχετε να μα προτείνετε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπιλμπά, παρακαλώ. Sí, muchas gracias, ministra, por Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και για τις εξηγήσει και για την προσήλωσή σας ε, στην πραγματική αποκατάσταση της ισότητας ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη με κάλυψαν ε, οι προλαλήσαντες σε πολλές από τις ερωτήσεις που μου ήρθαν στο μυαλό. Έχω μια τελευταία. Όταν μιλήσατε για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας, ε, μας φέρει στο μυαλό το γεγονός ότι η βία μεταξύ των φύλων είναι απόρρια της ανισότητας που υπάρχει μεταξύ των δύο φύλων. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας που προτείνεται περιλαμβάνει και τη δυνατότητα να εφαρμοστούν τα ίδια πρωτόκολλα δράσης μεταξύ των χωρών. Γιατί όπως ξέρετε η χώρα των Βάσκων ενέκρινε το 2005 το τον πρώτο νόμο στην Ισπανία για την ισότητα ανδρών γυναικών με πολύ προηγμένα μέτρα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της βίας μεταξύ των φύλων. Και επεξεργαστήκαμε ιδιαίτερα το θέμα των πρωτοκόλων δράσης, ώστε και τα υγειονομικά αλλά και τα αστυνομικά πρωτόκολλα στα δικαστήρια να είναι τα ίδια, ώστε να μπορεί να γίνει μια σύγκριση της κατάστασης. Αυτό λοιπόν το ευρωπαϊκό ένταλμα περιλαμβάνει αυτή τη δυνατότητα ομοιο γενοποίησης, ομοιομορφοποίησης ε, των πρωτοκόλων δράσης. Επίσης, ό,τι αφορά την εκστρατεία συνειδητοποίησης ή κοινωνικής αφύπνισης, δεν ε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια εκστρατεία με κοινό τους άνδρες. Στην χώρα των Βάσκων οργανώσαμε μια τέτοια εκστρατεία με τίτλο «Μεταξύ των ανδρών» ή για τους άνδρες με στόχο την πρόθεση ενός μανιφέστου υπέρ της ε, ισότητας. 10.000 βάσκοι, άνδρες βάσκοι, υπέγραψαν αυτό το μανιφέστο, αυτή τη διακήρυξη υπέρ της ισότητας. Δεν θα μπορούσαμε κάτι αντίστοιχο να το εφαρμόσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μία εκστρατεία συνειδητοποίηση που θα απευθύνεται στους άνδρες και θα έχει στόχο την προαγωγή της ισότητας μεταξύ των φύλων. Πιστεύω ότι ε, και στις εκθέσεις που γίνονται και στις φωτογραφίες που βλέπουμε και εδώ και στις εθνικές βουλές βλέπουμε ότι η εικόνα της εξουσίας έχει ανδρικό πρόσωπο. Φαίνεται ότι σε όλες τις εκστρατείες που γίνονται η φωτογραφία για την εντύπωση που δίνεται για το πρόσωπο της εξουσίας είναι πάντα ανδρική. Και εκεί λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια προσπάθεια. Στη χώρα των Βάσκων είχαμε επίσης ε, ε, το αξίωμα του διαμεσολαβητή για την ισότητα που επιλαμβανόταν των προσωπικών καταγγελιών που γινόταν από γυναίκες, των ιδιωτικών καταγγελιών. Γιατί σε θέματα δημόσιας διοίκησης δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για τις ιδιωτικές καταγγελίες δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στον οποίο θα μπορούσαν να αποταθούν οι γυναίκες. Στη χώρα των Βάσκων υπάρχει ένας ειδικό διαμεσολαβητής για θέματα ισότητας. Δεν θα μπορούσατε κάτι αντίστοιχο να το προτείνετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναν Ευρωπαίο διαμεσολαβητή για την ισότητα, ώστε και οι γυναίκε που εργάζονται σε ιδιωτικέ επιχειρήσει, στον ιδιωτικό κλάδο, να μπορούν να αποτείνονται σε κάποιον αρμόδιο και να μπορούν να κάνουν τι καταγγελίε του. Ευχαριστούμε κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Υπουργέ, και εγώ να σα καλωσορίσω και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Ισπανική Προεδρία. Τα θέματα ισότητα τα συζητούμε πολλά χρόνια και συνήθω οι διαγνώσει μα είναι πανομοιότυπε. Η δική μου ερώτηση είναι πιο πρακτική. Παρακολούθησα πριν μερικά χρόνια την πρωτοβουλία της Γερμανικής Προεδρίας, η οποία εισήγαγε το θεσμό του gender budgeting. Και διερωτούμε, η Ισπανική Προεδρία έχει πρόθεση να ακολουθήσει τέτοιου είδους καλές πρακτικές, ούτω ώστε να βρίσκονται πρακτικές λύσεις στην αντιμετώπιση προβλημάτων όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει κάνει πάρα πολύ ε, επιτυχημένη εκστρατεία του 2006-2008 με τη συνεργασία όλων των κοινοβουλίων για πρόληψη καταστολή της βίας. Διερωτούμε εάν ε, μπορεί να αξιοποιηθούν και τα reports και οι εμπειρίες του Συμβουλίου της Ευρώπης ούτως ώστε στο θεωρητικό μέρος εφόσον έχουμε πανομοιότυπες αντιλήψεις να πάρουμε τη διάγνωση ως δεδομένη και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να βρει συγκεκριμένε ολοκληρωμένε στρατηγικέ αντιμετώπιση να είναι πιο πρακτικό ο τρόπο με τον οποίο εμεί νομοθετούμε και βρίσκουμε στρατηγικέ για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. διαφορετικά αν μένουμε μόνο στη θεωρία θα συζητούμε για πολλά χρόνια και θα κάνουμε διαγνώσει χωρί πρακτικού τρόπου αντιμετώπιση. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να ακούσω πιο συγκεκριμένα πρακτικών τρόπων αντιμετώπιση και κυρίω εφαρμογή μεθόδων gender budgeting στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Μάλιστα, τώρα η κυρία Ματήρα, η αντιπρόεδρός μας. Ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. κύριε Υπουργέ. Παρότι θα σας ε, υποβάλω μια ερώτηση που έθεσε ήδη ο συνάδελφός μας, ο κύριος Ταραμπέλα, παρόλα αυτά θα την υποβάλω γιατί θέλω να επιμείνω στο θέμα, παρότι δεν είναι το μόνο. Λοιπόν, ε, τι, ποια είναι η άποψή σας για τη θεσμοθέτηση μια, ενός ευρωπαϊκού έτους για την βία κατά των γυναικών. Αναφερθήκατε ε, στις διασκέψεις που θα οργανώσετε. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναλυφθεί στην Ιταλία και στη Νέα Υόρκη. Οπότε, όπως και ο κύριος Ταραμπέλα, θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, διότι η παρουσία σας εδώ καταδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση που έχετε για τα θέματα που είναι το αντικείμενο εργασίας της Επιτροπής μας. Κυρία Ζαμπόφσκα τώρα. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Μια πολύ σύντομη και συγκεκριμένη ερώτηση. Ακούσαμε όλοι ότι είναι προς το συμφέρον ε, των πάντων να υιοθετήσουμε μια οδηγία για την ασφάλεια, την ασφαλή εργασία των εγγύων γυναικών. Αυτή η οδηγία ξέρουμε ότι συζητείται εδώ και πολύ καιρό. Κύριε Δεφορά, μεταξύ των ε, ε, πολιτικών ομάδων ήταν η θέση ως προς την ε, εισαγωγή μιας άδεια πατρικής. Εμείς συμφωνούμε από το ΕΛΚΟ ότι θα πρέπει ο πατέρας να συμβάλλει στην ανατροφή των παιδιών. Αλλά πιστεύουμε ότι το ζήτημα της πατρικής άδειας δεν έχει θέση μια τέτοια οδηγία και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από μια διαφορετική, από ένα διαφορετικό νομοθέτημα. Η Ισπανική Προεδρία λοιπόν τι στάση θα τηρήσει στη διαπραγματεύσει του Συμβούλιο. Ξέρω ότι δεν είναι ε, το ερώτημα που σας υποβάλλω και εύχομαι και κάθε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόφσκα. Η Υπουργό ε θα ξαναπάρει το λόγο για να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα που δείχνουν τη δέσμευση των μελών της Επιτροπής μας. Σα ευχαριστώ θερμά και πάλι για τι παρατηρήσει σα. Θα αρχίσω από την τελευταία παρατήρηση για την ισπανική θέση ότι αφορά την οδηγία για την άδεια μητρότητα. Αν και το είχα πει και στην αρχή. Προκειμένου να καταλήξουμε στη συμφωνία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να συνεννοηθούμε, να καταλήξουμε σε συνένεση και άρα να εγκρίνουμε αυτή την οδηγία. Αυτό είναι ο πρωταρχικός στόχος της Ισπανικής Προεδρίας. Πιστεύουμε ότι για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία θα πρέπει η οδηγία αυτή να είναι ισορροπημένη και να αντικατοπτρίζει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Θα πρέπει να βρεθεί ισορροπία μεταξύ της έντασης ε, των αποδοχών και της διάρκειας της άδεια. Φυσικά τα μέτρα αυτής της οδηγίας θα πρέπει να προωθούν την υγεία της μητέρας, θα πρέπει να προωθούν την ανάνυψη της μητέρας μετά το τοκετό, αλλά να αυξάνει και την ε, νομική ασφάλεια, αλλά και να διευκολύνει την επανένταξη στην αγορά εργασίας. θα πρέπει η γυναίκα μετά τον τοκετό να αντιμετωπίζει δυσκολίε στην επανένταξή τη στην αγορά εργασία. Επίση, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την οδηγία για να προαγάγουμε τη συμφιλίωση, το συνδυασμό του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο. Και όλα αυτά με μια ευρεία, με μια ελαστική προοπτική και φυσικά ασκώντα ε, μια συνυπευθυνότητα και προωθώντα ε, τον ισότιμο καταμερισμό των ε, οικογενειακών βαρών και καθηκόντων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ισπανική Προεδρία θα ενισχύσει τη συνεργασία τη και με το Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτύχει μια εναρμόνιση του επίπεδου προστασία για τι έγκυε, τι λεχόνε και τι γαλουχούσε γυναίκε. Πάντω, αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις ψηφοφορίες και τις εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις και της δικής σας Επιτροπής και της Επιτροπής Απασχόλησης και ανάλογα με την έκβαση αυτών των ψηφοφοριών θα προωθήσουμε το θέμα και την εναρμόνιση των θέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Όπως σας είπα αυτή είναι σημαντική προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας και πολύ θα θέλαμε να είχαμε ε, ξεκινήσει πιο νωρίς αυτό το έργο, αλλά από σεβασμό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίσαμε να περιμένουμε τις εκθέσεις και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις και ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι φορά το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, σας είπα με ρωτήσατε τι ακριβώς θέλουμε από το παρατηρητήριο. Δεν θέλουμε μια νέα δομή. Δεν θέλουμε ένα νέο οργανισμό ή μια νέα υπηρεσία, αλλά θέλουμε μια λειτουργική οργάνωση για να καταλήγουμε σε δείκτες, ε, σε εναρμόνιση μιας ε, μεθοδολογίας για τη συγκέντρωση των στοιχείων, ώστε να μπορούμε να καταλήγουμε σε συγκρίσιμα στοιχεία. Θέλουμε να καταρτήσουμε ένα κατάλογο των πρακτικών, να δούμε το θέμα της βίας μεταξύ των φύλων υπό το πρίσμα το υγειονομικό, αστυνομικό, δικαστικό, κοινωνικής προστασίας και όλα αυτά με τρόπο ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή τη γνώση στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να κάνουμε το πρώτο βήμα καταρτίζοντας κάποιους κοινούς δείκτες. Γιατί το πρόβλημά μας είναι κοινό, μαστίζει όλες τις ε, ευρωπαϊκές χώρες και κοινωνίες. Γι' αυτό και οι λύσεις ε, θα πρέπει να είναι κοινέ. Όταν τα προβλήματα είναι παγκόσμια, οι λύσεις παγκόσμιες. Όταν τα προβλήματα είναι κοινά και οι λύσεις θα πρέπει να είναι κοινέ. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στη διάθεσή μας ένα εργαλείο με στοιχεία, δείκτες, δεδομένα για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ομοιόμορφες πληροφορίες και εναρμονισμένες και να τις αξιοποιήσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Ταραμπέλα, το, το αρχικό σας σχόλιο με άφησε άναβη. μάλλον ως φιλοφρόνηση το εκλαμβάνω. Δεν θα επιμείνω σε αυτό. Επίσης, ε, ε, για την ερώτησή σας που την επανέλαβε και η κυρία Ματέρα, θα ήθελα να πω ότι για να θετήσουμε την απόφαση για το Δάφνη 2, Είπαμε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν από κοινού την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της βίας κατά των ε, κοριτσιών και γυναικών. Τα κάτι πιο συγκεκριμένο, όχι μόνο γενικά βία κατά των γυναικών. Φυσικά το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις στα πλαίσια των νομοθετικών αρμοδιοτήτων του, επί τη βάση όμως ε, του δικαιώματος της νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, μια και μας έχει μείνει ελάχιστο χρόνος, δεν θα ήθελα να αφήσω αναπάντητη καμία ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την παρουσία των γυναικών στα κέντρα λήψη αποφάσεων και σε ηγετικέ θέσεις, αυτό θα πρέπει να το δούμε όχι μόνο υπό το πρίσμα της δικαιοσύνης, που είναι και θέμα βέβαια δικαιοσύνης, αλλά είναι και θέμα αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα, αποδοτικότητα, παραγωγικότητα. Γιατί το 60% των πτυχιούχων ανατάτων σχολών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γυναίκες. Και μάλιστα τα βιογραφικά τους είναι πολύ πιο εντυπωσιακά από των ανδρών. Παρ' όλα αυτά, ούτε η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά είναι καλύτερη, ούτε η συμμετοχή τους ε, σε ηγετικές θέσεις είναι μεγαλύτερη, ούτε οι αμοιβέ τους καλύτερες. Και μάλιστα, μόνο 3% ε, των ε, ηγετικών θέσεων σε επιχειρήσεις σημαίνει στο χρηματιστήριο είναι γυναίκες. Ελάχιστες ε, είναι οι θέσεις του στα διοικητικά συμβούλια. Αυτό όχι μόνο είναι άδικο, αλλά είναι και αναποτελεσματικό. Γιατί δεν, δεν αξιοποιείται το τεράστιο δυναμικό που, συμπεριφ... που φέρουν οι γυναίκες. Και μάλιστα μία μελέτη λέει ότι οι γυναίκες σε ηγετικές, σε ηγετικές θέσεις δίνουν 43% μεγαλύτερη παραγωγικότητα, αποδοτικότητα στο επενδυμένο κεφάλαιο. Σίγουρα η συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις έχει ωφέλη σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Και αν θέλουμε μεγαλύτερη ενσωμάτωση και παρουσία των γυναικών στις ε, ηγετικές θέσεις, στις ηθήνουσε θέσεις, Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και δεν είναι μόνο απαραίτητο, αλλά είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό, όπως δείχνουν και οι μελέτες. Η προαγωγή της ισότητας είναι πολιτική αξία και της Ισπανικής Προεδρίας. Θα επιμείνουμε λοιπόν και στην καλύτερη παρουσία των γυναικών στις ηγετικές θέσεις, οικονομικές, πολιτικές, επιχειρηματικές και αυτό το θέμα θα το εντάξουμε και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020. Γι' αυτό και με... θα έχουμε και την κοινή πρωτοβουλία και το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ισότητας που θα γίνει το Φεβρουάριο στο Κάδη λίγες μέρες πριν από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το Πεκίνο σε 15 και θα συζητήσουμε κυρίως αυτό το θέμα προκειμένου να άρουμε τα εμπόδια στην πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και στην πρόσβαση και παραμονή τους στις ηγετικές και ηθήνωσες θέσεις πολιτικού, επιχειρηματικού και οικονομικού χαρακτήρα. Τέλος, να αναφερθώ και στα στερεότυπα. Κάποια ευρωβουλευτή το έθιξε. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το θέμα των στερεοτύπων θα το εξετάσουμε στις 31 Μαΐου σε μια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων στη Μαδρίτη. Εκεί θα αναφερθεί το θέμα των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και την πρόθεση της θέσης των γυναικών στα μέσα μαζική ενημέρωση και στην παιδεία. Αυτό θα είναι κέριο θέμα και για την Ουγγρική Προεδρία και πραγματικά είναι πολλά τα πλεονεκτήματα από το σύστημα του τρίου γιατί επιτρέπει στις τρεις προεδρίες να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρόγραμμα και να το προωθήσουν εξασφαλίζοντας μια συνέχεια που είναι πολύ σημαντική στους τομείς αυτούς. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό για θέματα ισότητα φύλων, το θέμα αυτό θα απασχολήσει το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργών Ισότητα που θα γίνει στη Βαλένθια. Γιατί και εκεί θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο, γιατί έχουμε την Ισπανική Προεδρία. Μετά το νόμο τη ισότητα, όλε οι συμφωνίε, νόμοι και νομοσχέδια έχουν μία μελέτη επιπτώσεων υπό το πρίσμα τη ισότητα των φύλων. Και το 2009 είχαμε για πρώτη φορά μελέτη επιπτώσεων ισότητας φύλων στον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να προχωρήσουμε σε θέματα πολιτικής ισότητας. Ο προπολογισμό ουσιαστικά περιλαμβάνει τις πολιτικές προτεραιότητες μιας κυβέρνησης και η συμπερίληψη της ισότητας των φύλων στις προτεραιότητες αυτές είναι χαρακτηριστική και δείχνει πόσο σημαντικό είναι να, προχωρήσουμε με πυγμή και αποφασιστικότητα και να επιδιώξουμε την ισότητα των φύλων, εφοδιάζοντας τον αγώνα μας με τα απαραίτητα οικονομικά μέσα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ΑΕΤΗΣ, γιατί τέθηκε μια ερώτηση σχετικά. Νομίζω ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις θα έχουμε τέτοια ευκαιρία να δείξουμε το ηθικό μας παράστημα ως Ευρωπαίοι και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σε μια τραγωδία τέτοιων διαστάσεων καλούμαστε όλοι να εκφράσουμε την προσήλωσή μας ε, προς τις αρχές μας, τη δέσμευσή μας ε, και τη αλληλεγγύη μας προς τις χώρες που πλήττονται περισσότερο. Γιατί ακόμη και στις χώρες αυτές οι γυναίκες πληρώνουν τα σπασμένα και είναι αυτές που φέρουν τη μεγαλύτερη οδύνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αναλάβει τη δέσμευση να βοηθήσει όσο μπορεί και θα φροντίσουμε ώστε να μπει στο δρόμο της αποκατάστασης το συντομότερο δυνατό η ΑΕΤ και μάλιστα γίνεται σχετική διάσκεψη και στο Μοντρεάλ γιατί έχουμε πολλά να συμβάλλουμε εδώ και θα παίξουμε πραγματικά το κύρος μας σε ό,τι αφορά τη στάση μας προς την αιτία. Για το παρόν και το μέλλον της. Ευχαριστώ. Ένα θερμό ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, γιατί δώσατε και διεξοδικές και σαφείς απαντήσεις. Δείχνετε ιδιαίτερη προσήλωση στα θέματα ισότητας. Εξ ονόματι της Επιτροπής θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ισπανική Προεδρία Ελπίζουμε να καταφέρει να προάγει όλα τα ζητήματα της ισότητας των δύο φύλων. Να θερμό ευχαριστώ και πάλι και καλή επιτυχία. Μάλιστα, συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο σημείο. Είχαμε προβλέψει οι ψηφοφορίε να αρχίσουν λίγο νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει γιατί ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτησή μα. Οπότε περνούμε στο σημείο 5, απαλλαγή για το 2008. Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Τμήμα 3, Επιτροπή. Η συγγήτρια της Επιτροπής μας είναι η κυρία Μπάουερ. Κυρία Μπάουερ, θέλετε να μας ενημερώσετε για οτιδήποτε πριν να αρχίσουν οι ψηφοφορίες ή να αρχίσουμε. Έχετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να σημειώσω πριν ξεκινήσουμε ότι δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίες και παρά αυτό να προσθέσω άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Είσαστε έτοιμοι συνάδελφοι για να αρχίσουμε. Για τον προϋπολογισμό. μπορούμε ομαδών να ψηφίσουμε όλες ε, τις ε, τροπολογίες, όλες τις παραγράφους. Υπάρχουν ενστάσεις, μπορούμε από κοινού να τα ψηφίσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Θα αρχίσουμε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω στα αγγλικά κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων για τα κακά μου αγγλικά ε, θα... και κάντε μου νόημα αν κάτι δεν καταλαβαίνετε και θα το εξηγήσω. The opinion, uh, Mrs. Powers, Η γνωμοδότηση της κυρίας Μπάουερ. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Ναι, ναι, έχουμε και τελική ψηφοφορία βεβαίω. Με τις κάρτες μας, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία, άρχεται. Θα περιμένουμε ένα λεπτάκι για να, ε, για να βρείτε την κάρτα σας. Ψήφισαν όλοι παρακαλώ. Everyone voted no. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίθηκε. 22 ψήφοι υπέρ. Ομόφωνα εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κυρία Μπάουερ. Το επόμενο σημείο για τις ψηφοφορίες μας είναι δύο προφορικές ερωτήσεις για το Πεκίνο ΣΥΝ 15. Σας ερωτώ, μπορούμε από κοινού να, τις, ε, να ψηφίσουμε για αυτές τις προφορικές ερωτήσεις ε, προς την Επιτροπή και προς το Συμβούλιο αντίστοιχα. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί, τις δύο ερωτήσεις. Ωραία. Υπέρ παρακαλώ. Amendment 7, excuse me. Ζητώ συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Ναι, δεν ψηφίζουμε για το ψήφισμα, για τις προφορικές ερωτήσεις ψηφίζουμε τώρα. Υπέρ παρακαλώ, υπέρ για τις προφορικές ερωτήσεις. Κατά, αποχές εγκρίνονται. And now we go to the resolution concerning Beijing plus 15. Πάμε στο ψήφισμα για το Πεκίνο συν 15. Περνάμε στην ψηφοφορία για το ψήφισμα. Τροπολογία 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές.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 Ψηφίστε παρακαλώ. 18, έτσι. Πέραση της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 23. 15 υπέρ. Σύνολο ψηφισάντων 23. 15 ψήφοι υπέρ. 8 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη επίση. The electronic vote. Ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 22 για εξακρίβωση. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας. 13 ψήφοι υπέρ, 12 κατά. Εγκρίθηκε τελικά. Η πρώτη τροπολογία υπέρ παρακαλώ κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 λέει η πρόεδρο. 4 διορθώνει τώρα. Όχι, υπέρ. Η τροπολογία 3 υπέρ. Διορθώνει τώρα η πρόεδρο. Η τροπολογία 4 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Απορρίφθηκε. Τώρα είναι η τροπολογία 3 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έξι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική για το σύνολο του ψηφίσματος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά τρεις αποχές. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους μας. Okay, då går vi till nästa Περνούμε στο επόμενο σημείο τώρα. som er, eh, Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2009. Ο κύριος Ταραμπέλα, ο εισηγητής μας, θα πάρει πρώτος το λόγο, παρακαλώ. Θα είμαι σύντομο. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα, έστω και αν ε, μας πήρε τόσο χρόνο με την ε, συνάδελφό μου με την βοηθό μου να ετοιμάσουμε αυτήν την ε, έκθεση. Θα ήθελα να είχαμε περισσότερο χρόνο επαφή, συνεδριάσεις. Μόνο τέσσερις μπορέσαμε να κάνουμε. Και με σύμπτωση χρονική των δύο εκθέσεων της κυρίας, με την κυρία Λούλινγκ ως κοιόδη πρέπει να πω ότι χρειάστηκε πολύ ενεργητικότητα από πλευράς μου να δουλέψω ιδιαίτερα για την άλλη έκθεση που αφορούσε τις, ε, τη σήμανση των προσυσκευασμένων τροφίμων στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να κάνουμε μια συνεδρίαση να τα πούμε, αλλά δεν ε, τα καταφέραμε. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδες συγκητές, όλους όσοι κατέθεσαν τροπολογίες, όσους ενδιαφέρθηκαν, και την, όσους ενδιαφέρθηκαν και την έκθεση. Ευχαριστώ κυρίως για το τόσο καλό κλίμα μέσα στο οποίο συνεργαστήκαμε. Απλώς θα σημειώσω ότι όπου δεν μπόρεσα να καταλήξω συμβαστική λύση, ας πάμε να ψηφίσουμε και με την ψηφοφορία να βγει ο καλύτερος. Ευχαριστούμε κύριε Ταραμπέλα. Δεν θα κάνουμε τώρα μακροσκελή συζήτηση, ελπίζω. Κάποιες μικρές παρεμβάσεις. Η κυρία Λούλινγκ θα πάρει πρώτη το λόγο. Πρόεδρε. Δεν ξέρω ποιος, ποιος απορρόφησε την ενέργεια Τίνος, την ενεργητικότητα Τίνος για την έκθεση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η έκθεση του κυρίου Ταραμπέλα είναι πολύ σημαντική έκθεση. Και πιστεύω ως εκ τούτου ότι θα πρέπει να μην την καταστήσουμε δυσανάγνωστη με την εισαγωγή διαφόρων αιτιολογικών σκέψεων και λοιπόν παραγράφων οι οποίες δεν μας βρίσκουν αντίθετους αλλά που ε, βαραίνουν τόσο πολύ το κείμενο σε βαθμό που να το καθιστούν δυσανάγνωστο. Για να μην μιλήσω για εκείνους οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία ε, προσθέτουν και άλλες λεπτομέρειες και παρατηρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Και έχω κάνει και τον κατάλογο των ψηφοφοριών για την ομάδα, τόσο από τους συναδέλφους να αποσύρουν δικές τους τροπολογίες, συναδέλφους από την ομάδα μου, να αποσύρουν τροπολογίες τις οποίες θεωρώ μη ουσιώδους σημασίας σε μια έκθεση όπως η δική σας η οποία μου φαίνεται ότι θα πρέπει να εστιάσετε στο ουσιοδέστατο και να παραμένει ευανάγνωστη. Γι' αυτό έχουμε ένα τέτοιο κλιμακωτό θα έλεγα κατάλογο ψηφοφοριών. Για το καλό του κυρίου Ταραμπέλα το κάναμε. Για να μην φορτωθεί, για να μην παραφορτωθεί αυτή η έκθεση. Γιατί ξέρετε πολύ συχνά παραφορτωμένες μαούνες βουλιάζουν. Ευχαριστούμε κυρία Λούλιν. Κυρία Ζαμπόσκα, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αποσύρω την τροπολογία παριθμών 44 διότι ανήκει ουσιαστικά στην έκθεση για την αντιμετωπίση των διακρίσεων ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών και μεταξύ γενναίων και λεγγύης μεταξύ γενναίων. Από Σύρο λοιπόν τροπολογία παριθμών 44. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γιάννα Κουδάκη τώρα παρακαλώ. Η κυρία Γιάννα Κουδάκη, ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση και νομίζω συμφωνούν όλοι. Δηλαδή, η σημίστη η κατάργηση διακριτική μεταχείριση στον χώρο εργασία, η ισότητα των δύο φύλων, ε, φυσικά, όπω και οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε, μα είναι ιδιαίτερα προσφυλή αυτά τα θέματα. Όμω, όπω πάντα, όταν μιλάμε για αναπαραγωγική υγεία με στην έκθεση, ε, δεν είναι αρμόζον. Είναι θέμα ε, εθνικό αυτό και όχι ευρωπαϊκό. Ε, τώρα, μιλώντας για αναπαραγωγική και αναπαραγωγική υγεία, τι κάνουμε, νερώνουμε την έκθεση και υποβαθμίζουμε άλλα σημαντικά ζητήματα, τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των μισθών, σαν ευχολόγιο είναι, που τελικά όμως ε, θα υπογράψει την καταδίκη μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα αναφέρουμε όλα αυτά. Μάλιστα, η κυρία Κορνέλισον. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά σημειώνω ότι είναι πολύ ευχάριστο να συζητάμε τέτοια θέματα με τόσο ευηδή εισηγητή. Όχι, κοροϊδεύω, λέει η κυρία Κορνέλισαν. Πολύ καλή λοιπόν και πληρέστατη αρχική έκθεση. Ίσως παρά ήταν περιεκτική, αλλά αυτή είναι και η φύση μιας έκθεσης αξιολόγησης. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε κάπως πιο οξυμένες ή πιο σαφείς διατυπώσεις και αυτό προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε κάποιες τροπολογίες που έχουμε καταθέσει και θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα πολύ σύντομα. Καταρχάς, ε, σχέδια αποκατάσταση αποκρίσεις ή αντιμετώπισης. Λυπούμε που απέρριψε την υπαριθμό 46 τροπολογία μου εισηγητής γιατί αναφέρεται στο γεγονός ότι τα σχέδια για οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών επικεντρώνουν, συγκεντρώνονται λίγο πολύ σε τομείς όπου κυριαρχούν οι άνδρες. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα και 90% των κονδυλίων του ταμείου αυτού το εισπράττουν άνδρες το πολύ 10% πάει σε γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας άνδρας ο οποίος έχει χάσει τη θέση εργασία του θα πρέπει να μην ε, ε, λάβει την κατάλληλη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρέπει και να είμαστε διατεθειμένοι, χάρη στην κρίση και τις ευκαιρίες που προσφέρει, αν δούμε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική, να προσφέρουμε βοήθεια στοχευμένη στις γυναίκες και ελπίζω ο εισηγητής να υποστηρίξει την υπαριθμό 46 τροπολογία μου. Επίσης, οι γυναίκες στην λήψη αποφάσεων. Με έκπληξη βλέπω πάντοτε ότι ναι, όλα τα κόμματα το βρίσκουν πολύ σημαντικό το θέμα. Μεν, πλην όμω δεν είναι όλα διτεθειμένα να προβούν ε, σε μέτρα που θα προωθούσαν περισσότερο το θέμα αυτό. Εγώ από 17 ετών αγωνίζομαι για τα δικαιώματα της γυναίκας. Έχουν περάσει έκτοτε 20 χρόνια. Το θέμα παραμένει ανεπίλητο και μόνο η Νορβηγία έχει να επιδείξει πραγματικές πρόοδους. Και ασφαλώς θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Συχνά προβάλλεται ως ε, ε, επιχειρήμα το γεγονός ότι είναι προσβολή για τη γυναίκα να την στηρίξουμε ή ότι δεν είναι ε, ισότιμος ο ανταγωνισμός, δεν είναι δίκαιο εγώ θα έλεγα δίκαιο δεν μπορεί να είναι ποτέ όσο οι συνθήκες είναι αρνητικές εις βάρος των γυναικών. Και για παράδειγμα θα σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν ε, σε μια συνεδρίαση με ε, αρχηγούς, με διευθυντές επιχειρήσεων σε, ε, στη σύνταξη μάλιστα οι οποίοι μου ζήτησαν ε, να του σερβίρω τον καφέ, γιατί θεώρησαν ότι για να είμαι γυναίκα μάλλον ε, προέρχομαι από το χώρο της εστίαση ε, και, και το καφενείο. Αυτό λοιπόν, μέχρι να αλλάξει αυτή η νοοτροπία δεν έχουμε κάνει τίποτα για τα δικαιώματα της γυναίκας. Επίση, θα ήθελα να υποστηρίξω την τροπολογία υπαριθμών 91 τη ΑΛΔΕ, χωρί όμω να καταλαβαίνω ταυτόχρονα και γιατί δεν συμφωνεί η ΑΛΔΕ από πλευρά τη για ένα χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών. Καταλαβαίνω ότι το ΕΛΚ δεν θα ήθελε ένα τέτοιο χάρτη, αλλά η ΑΛΔΕ γιατί να μην, έχει, να μην δεχθεί μέσα ειδικά ε, για την εξασφάλιση τη ισότητα ανδρών και γυναικών. Και αν υπάρχει κάποιο από την ε, ομάδα των φιλελευθέρων, παρακαλώ να μου εξηγήσει περισσότερο την ε, άρνηση αυτή. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ταραμπέλα για τα, τις καταλεκτικές παρατηρήσεις του. Υποθέτω ότι η κυρία Κορνέλισεν ε, στη συνάντηση που προανέφερε τελικά δεν τους έρβηρε τον καφέ έτσι. ελπίζω να σηκώθηκαν μόνοι τους να τον πάρουν τον καφέ τους έτσι είμαι πεπισμένη Κύριε Ταραμπέλα παρακαλώ να ευχαριστήσω τις συναδελφούς για τη συνδρομή τους. Ας περάσουμε στο ψαχνό. Τροπολογίες 94 της κυρίας Κορνέλσεν και 91 της κυρίας Ινβέλτε. Μα είχα ταχθεί ήδη υπέρ. Σας ε, καθησυχάζω ε, για την... Ε, για τις 46 έχουμε πιέσει από συναδέλφους, αλλά ε, ζούμε μέσα σε μια πραγματική οικονομία. Αν θέλουμε να ξεκινήσει και πάλι η ατμομηχανή της οικονομίας, Υπάρχουν αυτά τα φαλοκρατικά στερεότυπα που πρέπει να καταπολεμήσουμε, ναι μεν, αλλά η πραγματικότητα παρότι μπορεί να είναι πράσινη, νέα, μιλάμε για δημόσια έργα, για ευρωπαϊκούς υδροδρόμους, ε, η πλειοψηφία άντρες θα είναι. Και ήταν και τα πρώτα θύματα, γιατί στη βαριά βιομηχανία σημειώθηκαν οι πρώτες απώλειες θέσεων απασχόλησης και φυσικά έπεσαν θύματα και οι γυναίκες, γιατί με διαδοχικά δήματα, ε, κύματα συγγνώμη, επηρεάστηκαν και οι δημόσιες υπηρεσίες, όπου συνήθως ως επιτοπλίστων εργάζονται οι γυναίκες. Για τις κοινωνικές υπηρεσίες, ναι μεν, ναι, να τα κάνουμε όλα αυτά που λέμε, αλλά πρώτα να ξεκινήσει η πραγματική οικονομική ατμομηχανή. Ε, λέμε εδώ ότι αν ανάκαμψη τη οικονομία. Λυπούμεθα που η ανάκαμψη τη οικονομία βασίζεται σε επαγγέλματα που ανδροκρατούνται. Ναι, ναι, το δέχομαι, δεν το αρνούμε, αλλά είναι απαραίτητο να επενδύσουμε σε αυτού του τομεί όπου σημειώνεται πλειοψηφία ανδρών. Γιατί αυτό επιβάλλει οικονομική πραγματικότητα. Σε έναν ιδανικό κόσμο, ναι, θα βρίσκαμε θερμοκολήτριε ε, ε, στον ίδιο αριθμό με του θερμοκολλητές. Αλλά τι θα κάνουμε. Στον ιδανικό ε, κόσμο θα ε, ενέκρινα την τροπολογία. Εντάξει, αν επιμένετε να την υποστηρίξω την τροπολογία, αλλά είχα ταχθεί κατά γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και έρχομαστε αντιμέτωποι με αυτή την πραγματικότητα που σας εξήγησα. Ευχαριστούμε κύριε Ταραμπέλα. Υπάρχουν άλλα σχόλια κυρία Φιγκυρέιντου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είχα ζητήσει αρχικά το λόγο, αλλά ακούγοντας τώρα αυτή τη συζήτηση σκέφτηκα να ζητήσω το λόγο, διότι ενώ είναι αλήθεια ότι στην πρώτη φάση απολέστηκαν περισσότερες θέσεις εργασίας στους ανδροκρατούμενους τομείς, ε, αυτό δεν ισχύει παρόλα αυτά τώρα. Τα τελευταία δεδομένα της Eurostat καταδεικνύουν ήδη ότι οι γυναίκες έχουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Συνεπώς ε, είναι πολύ λογική αυτή η τροπολογία για να αποδοθεί ιδέως αβαρύτητα σε αυτό το θέμα. Πέραν του όμως Υπάρχουν χώρες όπου το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι κατά πολύ υψηλότερο. Δεν μιλώ για αριθμό ανέργων, έτσι, ε, γιατί υπάρχουν περισσότεροι άντρες στον ενεργό πληθυσμό, άρα έχουν έχουμε περισσότερους άντρες άνεργους, αλλά εγώ σας μιλώ εδώ για ποσοστό ανεργίας και υπάρχουν χώρες όπου η ανεργία είναι υψηλότερη στις γυναίκες, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχουν τα πράγματα, στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό ήδη έχουμε εισέλθει επανέλθει σε αυτή την κατάσταση που σα είπα. Παρότι στην αρχή ήταν σε ανδροκρατούμενου τομεί. τώρα όμω έχουμε εισέλθει σε άλλη φάση. Ευχαριστώ. Μάλιστα και ένα σχόλιο από την κυρία Γκουμάη. Θα ήθελα απλώ να καταφύσω σαφέ το εξή. το πρώτο κομμάτι της κρίσης, η πρώτη περίοδος κρίσης οφειλόταν και στα αυτοκίνητα και στον ε, κατασκευαστικό τομέα. Ε, οι άντρε ήταν αυτοί που έχασαν προ τη θέση εργασία του ω συνέπεια τη κρίση στην πρώτη φάση τη. Όμω αυτό ήταν λίγο πολύ ε, ένα παραπέτασμα, ε, γιατί στη συνέχεια άρχισαν να χάσουν, να χάνουν τις εργασίες τους οι γυναίκες και για αυτές δεν υπάρχει αρκετή στήριξη ή δυνατότητα επανεισόδου στην αγορά εργασίας και γι' αυτό αυτό το προπέτασμα θα θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα που αφορούν τις γυναίκες με το Ταμείο. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συζήτηση και αρχίζουμε την ψηφοφορία, παρακαλώ. Ναι, ναι, θα ψηφίσουμε αυτό, είπαμε όλες. 45, ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται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 απορρίπτεται, τότε θα εξακριβώσουμε επαλήθευση ηλεκτρονική για την 68 παρακαλώ. Ψηφίστε 68, ψηφίστε με την κάρτα. Πέρας. Αποτέλεσμα 12 υπέρ, 15 κατά ότος, ότος απερίφθη. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 Είναι ταυτόσιμε αυτέ οι τροπολογίε Ομαδών παρακαλώ ψηφίστε από την 72 έω και την 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθησαν. 77. Δεν πρέπει να την ψηφίσουμε. Αναφέρεται not to be voted. 78. Σε δύο τμήματα παρακαλώ. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Αλλά ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 78. Ψηφίστε παρακαλώ. παρακαλώ. vote is closed. 12 voted for, 15 against. So... 12 υπέρ, 15 κατά, περίφθη. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 τώρα Α, καταπίπτει. Ογδόντα έξι. For. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 90 κατά τμήματα δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95, 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 91. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote Τέλος ψηφοφορίας. 27 ψήφισαν με 15 ψήφους υπέρ και 12 κατά. Εγκρίνεται. Η 96 καταπίπτει. 97. Απορι... Αποσύρεται. 98. Σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 100. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104. Ποιο είναι υπέρ. καταπίπτει λέει η πρόεδρος. 104. Λάθος διορθώνει. 104. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Η 103 καταπίπτει. Πάμε στην 105. ποιο είναι υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 106. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 7 και 8 και 9. Γιατί είναι επανομοιότυπες οι τρεις τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για τις τροπολογίες 107, 8 και 9. Άρχεται η ψηφοφορία. vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Έχει, έχει απορριφθεί. Απορριφθούν οι τρεις με 7 ψήφους υπέρ και 18 κατά. Μία αποχή. Οι 107, 108 και 109 απορρίπτονται. Τροπολογία 110. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 110 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote Τέλος ψηφοφορίας. Τώρα τελείωσε η ψηφοφορία. 9 ψήφισαν υπέρ, 14 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται η 110. Τροπολογία 111. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα δεν θα ψηφιστεί. Δύο. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ξεχωριστή ψηφοφορία για το, το θεωρώντας 8. Ποιος είναι υπέρ κατά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 Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. εποχές, Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. εποχές, Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Πρώτα υπέρ μάλλον λέει πρόεδρος. Ξανά, ξανά. Πρώτα, πρώτα υπέρ και μετά κατά. Υπέρ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Οι 14... 14 και 15 καταπίπτουν. Θα ψηφίσουμε την 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 18 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απόχες απορρίπτεται. Ή μάλλον να το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για την τροπολογία 21, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 13 ψήφισαν υπέρ και 14 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατάλληλη πρόεδρος πάλι πρώτα. Ε, συγγνώμη. Υπέρ. Υπέρ. Υπέρ, συγγνώμη, σας το συγγνώμη λέει η Πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 24, υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. 25, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. 26, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. ...27-28 καταπίπτουν. Τροπολογία 29 τώρα. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Ή... Δεν καταπίπτει, απλώς θα προσθεθεί. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε. Για την 29. Υπέρ, υπέρ της 29, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ως προσθήκη. Τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος κατά άποχες απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 ποιος είναι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 κατά πίπτη, συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, ε, κατά πίπτη συγγνώμη, 37, 38 και 39 μαζί γιατί είναι παρόμοιες. Ποιος είναι υπέρ, κατά άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον για τη 41. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. And nine voted for and 15 against. 9 υπέρ, 15 κατά και 3 αποχές. Απορρίπτεται λοιπόν η 41. 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Against. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 44 έχει αποσύρθει, οπότε τελική ψηφοφορία για το ψήφισμα με ηλεκτρονικό τρόπο άρχεται η ψηφοφορία. The vote Τέλος ψηφοφορίας. Ψήφισαν 15 υπέρ, 5 κατά και 7 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Ταραμπέλα. Συγχαρητήρια σε όλους μας βέβαια και στην Επιτροπή Σύσσωμη. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας στην ψηφοφορία. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 9 της ημέρας της διάταξης. Έχουμε την έκθεση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη δράση κατά του καρκίνου, Ευρωπαϊκή Σύμπραξη. Επί της ουσίας, αρμόδια είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σήμερα θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων και η συγκήτρια για την γνωμοδότηση, συντάξει γνωμοδότηση δηλαδή, είναι η κυρία Τόμψεν. Παρακαλώ κυρία Τόμψεν, έχετε το λόγο. Varsågod, φρου Thompson. μισής Thompson. Κυρία Τόμψεν, παρακαλώ. Κυρία Τόμψεν. I think it's very good you are so engaged, but the floor... Καλό είναι να κάνετε και την κουβέντα σας, αλλά το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε την έκθεση για τον ε, καρκίνο στην Ευρώπη και είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα διότι ο καρκίνος είναι μια πολύ σοβαρή απειλή κατά των ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως είναι διαφορετικοί οι τύποι καρκίνου που εμφανίζονται σε άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες κυρίως πλήττονται από ενδομήτριο, ε, καρκίνο, καρκίνο του τραχύλου της ε, μήτρας ε, και καρκίνο του μαστού. Ιδιαίτερα βλέπουμε να αυξάνονται τα ποσοστά των κρουσμάτων και ο καρκίνος να χτυπάει όλο και πιο νέες γυναίκες. 275.000 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση νοσούν από καρκίνο κάθε χρόνο. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εταιρική σχέση που βρίσκω ογκώδη και ενδιαφέρουσα υπάρχουν κάποιες πτυχές της ε, ε, προσέγγισης με βάση το φύλλο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των καρκίνων, την πρόληψη καλύτερα, που όμως δεν αναφέρονται όπως οι παραδείγματοι την ε, δυνατότητα, η δυνατότητα της έγκαιρης ανείχνευσης, ανείχνευσης των ε, καρκίνων των, στις γυναίκες ε, μαστού τραχύλου της μήτρας είναι δυνατό να γίνονται και πρέπει να προωθηθούν τα προληπτικά αυτά εξεταστικά, εξεταστικές αυτές μέθοδοι η ανείχνευση αυτή αν θέλουμε να μειώσουμε το, τα κρίσματα καρκίνου. Εξετάσουμε τη συχνότητα εμφάνιση ορισμένων καρκίνων σε σχέση με το, γεν, με το φύλλο και να γίνει μια ειδική μελέτη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμσον. Κυρία Λεωτά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ την κυρία Τόμψεν. Είναι πολύ καλό το σχέδιό της. Σύντομο, 1500 στοιχεία μόνο έχει το κείμενο. Θα συμφωνήσω, τυπογραφικά στοιχεία. Θα συμφωνήσω λοιπόν, θα ήθελα απλώς κάποια σημεία να συμπεριληφθούν, ίσως να τα προτείνω με τροπολογία όσον αφορά την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση για τις γυναίκες μετανάστες. Γιατί και εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές, έντονες διαφορές μεταξύ διαφορών ε, τύπων καρκίνων. Ορισμένοι τύποι καρκίνων εμφανίζονται στις ε, μετανάστηδες, όπως ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, που είναι πολύ πιο συνηθισμένος σε Γυναίκε καταγόμενε από την Ινδία ή την Κίνα. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη. επιση την πρόληψη θα πρέπει να την κοιτάξουμε και σε σχέση με την ηλικία, στι πιο ηλικιωμένε γυναίκε. Ξέρουμε ότι γυράσκει ο πληθυσμό μα ότι αυξάνεται η ηλικία των πολιτών μα και ο καρκίνο εμφανίζεται και στις ηλικιωμένες γυναίκες με περισσότερη συχνότητα. Στην πρόληψη λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ιδέα για ε, έγκαιρη ανείχνευση και στις ηλικιωμένε γυναίκες. Επίσης, θα πρέπει να δούμε την πτυχή των θρησκευτικών ομάδων. Υπάρχουν ομάδες θρησκευτικές ή πολίτες προερχόμενοι από συγκεκριμένους θρησκευτικούς χώρους στους, από τους οποίους δεν προβλέπεται ή δεν προτείνεται η δυνατότητα της έγκαιρης ανείχνευσης για τις γυναίκες. Ένα παράδειγμα είναι η Μάλτα που δεν έχει τις δυνατότητες. Ε, έγκαιρη διάγνωση επίσης σημαίνει από τις μελέτες που έχουμε δει την ε, μελέτη και των παρενεργειών που ενδεχομένω έχουν οι μέθοδοι διάγνωση, οι διαγνωστικέ μέθοδοι, μερικέ φορέ φέρνουν αναγκαία και άλλα δευτερεύοντα ενδεχομένω προβλήματα. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη όταν προτείνουμε μια διαγνωστική μέθοδο. Μια νέα μέθοδος πρόληψης του καρκίνου φαρμακευτική μέθοδος μπορεί να είναι πάρα πολύ ακριβή επίσης και είναι απαράδεκτο την πρόσβαση να την έχει μόνο κάποιος εύρωστος οικονομικά. Γι' αυτό λοιπόν όταν μέγα τμήμα του γυναικείου πληθυσμού πλήττεται από τη φτώχεια, πολύ περισσότερο από ότι άντρε αντίστοιχα, ε, δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουν από αυτό το φαυλοκύκλο κύκλο της φτώχειας οι γυναίκες εάν ε, εκτός των άλλων και τα φάρμακα που χρειάζονται είναι τόσο ακριβά. Πρέπει και αυτό το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε κυρία Λέωτα. Η κυρία Παλιαντέλη τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, μια ερώτηση περισσότερο στην ε, συντάκτρια. Ε, προβλέπετε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής, στην ανακοίνωση της Επιτροπής ε, κάτι που να έχει σχέση με την έρευνα ή απλώς με διαπιστώσεις και αν σκέφτεται μια ευρωπαϊκή, ε, ανεξάρτητα από το φύλλο, μια υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των ε, Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Οβίρς τώρα. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι αξιόλογη. Και χαίρομαι ιδιαίτερω που αναλάβε η κυρία Τόμσεν τη Επιτροπή μα τη σύνταξη τη σχετική γνωμοδότηση. Εδώ ιδιαίτερω εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, έμφαση που δίνεται στους λόγους ε, ανάπτυξης των καρκίνων ε, η εμφάνιση των καρκίνων, αλλά νομίζω ότι και στην ενημέρωση, συνειδητοποίηση, εκστρατεία για την πρόληψη Μία λέξη κλειδί από την ανακοίνωση της Επιτροπής είναι η εταιρική σχέση. Η εταιρική σχέση σημαίνει ότι πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και άτομα φυσικά να εμπλακούν τόσο οι ενώσεις των ασθενών όσο και οι ιατροί, οι ιατρικοί σύλλογοι κτλ. Όταν δεν μιλούμε για προσβασιμότητα σε πληροφορίες σχετικές με τις θεραπευτικές αγωγές ή με την πρόληψη πολλές φορές διαπιστώνουμε σημαντικές διαφορές στι δυνατότητε που προσφέρονται σε κάθε κράτο μέλο. Πριν όμω πρέπει κάθε γυναίκα να έχει τη δυνατότητα τη πρόσβαση και στην ε, γνώση, τη σχετική, στην πληροφόρηση, τη σχετική με την πρόληψη, όσο και με την ε, θεραπευτική αγωγή. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο κείμενο λοιπόν. Για το 2013 και το και τις διαγνωστικές ε, μεθόδους, τα διαγνωστικά συστήματα που προτείνονται. Ε, ναι, βεβαίω, είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πολύ ρεαλιστική. Α είμαστε ρεαλιστικοί σε αυτά που ζητούμε, γιατί με δεδομένη την οικονομική κρίση θα πρέπει και να διαρωτηθούμε αν τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή εντό τριών ετών και δι' όταν του προσδιορίζουμε και χρονικό όριο το 2013. για τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Έτσι λοιπόν ίσως μια ή λεπτομερέστερη στρατηγική θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί για το τόσο αυτό ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τόμψεν τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Όβιερ, για να ξεκινήσω το τέλος. Ο στόχος μου είναι να αποφύγουμε τους θανάτους από καρκίνο των γυναικών. 275.000 το χρόνο είναι οι γυναίκες που νοσούν στην Ευρώπη από καρκίνο. Ε, κάτι πρέπει να κάνουμε λοιπόν γι' αυτό. Εγώ από τη Δανία έχω την εμπειρία ότι το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ή δυνατότητες που προσφέρονται μέσα σε ένα κράτος σε σχέση με ένα άλλο κράτος. Ακόμη και στην περιφέρεια ε, από τη μια περιφέρεια στην άλλη του ίδιου κράτου βλέπουμε διαφορέ. Υπάρχουν, χώρε, ε, ε, υπάρχουν περιοχέ στι οποίε δεν έχουν τη δυνατότητα του προσυμπτωματικού ελέγχου. Ε, Πώ θα γίνει, δεν θα πρέπει να πάει αυτή η γυναίκα κάπου να μεταβεί στην πρωτεύουσα σε μια κεντρική πόλη για να υποβληθεί σε αυτόν τον έλεγχο. Προφανώ για άλλη γυναίκα είναι πιο εύκολα τα πράγματα και για άλλη πιο δύσκολα στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Περιφερειακά έστω πρέπει κάτι να γίνει, να οργανωθεί κάποιο σύστημα και να διευκολύνουμε την πρόσβαση αυτή στον, στον προσυμπτωματικό έλεγχο, γιατί διαφορετικά δεν θα έρχονται οι γυναίκε. Καν δεν θα προβαίνουν σε αυτόν τον έλεγχο. Επίσης θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει οι οργανώσεις ε, νόσης προσώπων ή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια και την έρευνα. Εάν υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες η Επιτροπή θα πρέπει και εμείς να τις ε, στηρίξουμε. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά μέσα που θα επέτρεπαν ενδεχομένω και εμπλοκή τη αγοράς, αγορά εργασία ε, και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύσκολο όταν μια γυναίκα είναι ε, ήδη ασθενή, όταν έχει ήδη νοσήσει, είναι δύσκολο να προχωρήσει ε, ή σε εξέβρεση ε, εργασίας ή στην, ε, στα δεδρομία της ή επίσης ε, το ζήτημα με τις γυναίκες μετανάστες ή τα φαινόμενα ε, ε, ενδεχομένως γενετικών ή κληρονομικών καρκίνων που εμφανίζονται σε γυναίκες από την Ινδία, την Κίνα ή τη Λατινική Αμερική. Ίσως αυτό θα έπρεπε να το δούμε κάπως διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ζαμπόσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και το συγγνώμη που λαμβάνω το λόγο μετά την εισηγητρία που είχε ολοκληρώσει τι απαντήσει αλλά ήθελα ένα-δύο πράγματα να επισημάνω. Ίσως σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν όχι μόνο την έρευνα αλλά και την πρόληψη και την αγωγή και θεραπεία. Μιλάμε για οικονομική κρίση και λέμε ότι δεν έχουν τα κράτη στη θέση τους αρκετά κονδύλια. για τον τομέα αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσδιορίσει σαφείς στόχους. Στόχους για τους οποίους θα διαθέσει και τα κονδύλια που χρειάζονται. Και τα πολέμηση του καρκίνου νομίζω ότι πρέπει να είναι μια από τις προτεραιότητες. Κυρία Συγκητρία. Ε, είπατε και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει ανάγκη και περισσότερη έρευνα σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ καρκίνου και φύλου στο σημείο παριθμών 1. Ναι, συμφωνώ, αλλά ίσως θα έπρεπε να δώσουμε και πιο συγκεκριμένο χαρακτηρισμό στους, ε, στις αιτίες του καρκίνου. Να μην μιλάμε δηλαδή γενικά για τις επικίνδυνες ουσίες και τις επιπτώσεις του στη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. Είναι πολύ γενικόλογη αυτή η διατύπωση. Και δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών της Ευρώπης γιατί δεν θα τους εγγίξει αυτή η ε, διατύπωση. Εάν λοιπόν περιγράψουμε συγκεκριμένα τους λόγους, τις αιτίε καλύτερα, θα βοηθήσουμε πιστεύω τους πολίτες μας να συμπράξουν στην πρόληψη. έχοντας γνώση του ποιες είναι οι ουσίες οι οποίες μπορεί να έχουν επίδραση στην ε, υγεία τους. Ευχαριστούμε και θα ακούσουμε την κυρία Τόμψεν για να κάνει τα τελικά σχόλια. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω με την κυρία Ζαμπόρσκα για τα κονδύλια που χρειάζονται για την πρόληψη και την αγωγή, τη θεραπευτική αγωγή. Ε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε μια μορφή αρρώστηση η οποία πολλές φορές οδηγεί και σε απουσία μακροχρόνια από, την, από το χώρο εργασία, η οποία προκαλεί επιπλέον κόστος, κοστίζει δηλαδή περισσότερο στην κοινωνία. Επίσης ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον με την όψιμη τεκνογωνία η οποία μάλλον συνδέεται και με τον καρκίνο του μαστού. Γι' αυτό θα έπρεπε οι γυναίκες νωρίτερα να κάνουν παιδιά. Ευχαριστούμε. Ας δούμε τώρα το χρονοδιάγραμμα. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών είναι η Δευτέρα Φεβρουαρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 23 Φεβρουαρίου. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 16 Μαρτίου ψηφοφορία και η Ολομέλεια θα ψηφίσει τον Απρίλιο. Ε, μπορούμε να εγκρίνουμε το χρονοδιάγραμμα. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Το επόμενο σημείο τώρα. Στρέφομαι προς την κυρία Εστρέλα. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες για την έκθεση της κυρίας Εστρέλα για την οδηγία, για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας, για τις ε, μισθωτές που έγκυες, ελεχώνες και γαλουχούσες. Έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας. Ε, θα το θυμάστε σίγουρα ότι αναπέμφθηκε το θέμα στην Επιτροπή μας από την Ολομέλεια ε, τον Ιούλιο του 2009 συγκεκριμένα και η κυρία Εστρέλα και αποφασίσαμε μάλλον να ορίσουμε την κυρία Εστρέλα για να επιληφθεί τη συνέχεια των εργασιών και έχουν υποβληθεί τροπολογίες, σε αυτό το στάδιο έχουμε φτάσει. Έχουν μεταφραστεί δε σε όλες τις γλώσσες οι τροπολογίες και μπορούμε σήμερα να τις συζητήσουμε. Θα αρχίσουμε τη συζήτηση ακούγοντας την αντιπρόεδρό μας, την κυρία Εστρέλα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι πρώτη συζήτηση στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την πρότασή μου αυτή και θα συζητήσουμε σήμερα τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από ευρωβουλευτές και διάφορες πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεισφορά όλων σας. Κατατέθηκαν 169 τροπολογίες. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, κάτι που δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον των βουλευτών για αυτή την οδηγία και την ε, αθρώα συμμετοχή στη διαμόρφωση της έκθεσης. Ορισμένες τροπολογίες επαναλαμβάνονται ή είναι ταυτόσιμες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να διαμορφώσουμε κάποιες συμβαστικές λύσεις και να ομαδοποιήσουμε ορισμένες τροπολογίες. Αυτή είναι η δική μου επιθυμία τουλάχιστον και αυτή και αυτό είναι και το στίχημα που έχουμε να αναλάβουμε όλοι, να συνεργαστούμε στενά με τους και ηγητές, με τις πολιτικές ομάδες, για να καταλήξουμε σε μια ευρεία, όσο το δυνατό πιο ευρεία συνένεση γίνεται. Η οδηγία αυτή είναι άκρο σημαντική, έχει κέρια σημασία και όλους μας ενδιαφέρει να διεκπαιρεώσουμε τη διαδικασία αυτή το συντομότερο δυνατόν. Και μάλιστα έχω επίγνωση των κολλημάτων που αντιμετωπίζουμε και των εμποδίων που καλούμαστε να υπερκεράσουμε. Επαναλαμβάνω, δική μου επιθυμία είναι να καταλήξουμε σε ευρεία συνένεση και να καταθέσουμε στην Ολομέλεια μια σύγχρονη πρόταση, μια πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων γυναικών, στις ανάγκες των Ευρωπαϊκών οικογενειών και θα λαμβάνει ταυτόχρονα υπόψη τα βασικά συμφέροντα των παιδιών. Η δική μου στάση είναι ιδιαίτερα διαλλακτική και ελαστική. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που σε καμία περίπτωση δεν θα τις δεχτώ. Οι προτάσεις για παράδειγμα και οι τροπολογίες που ζητούν την κατάργηση της νομικής βάσης και το άρθρο 141 της συνθήκης για μένα είναι παράδειγμα, Γιατί η αφαίρεση αυτού του άρθρου από την νομική βάση θα σήμαινε απαράδεκτη οπισθοχώρηση και παλιδρόμηση σε σχέση με την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που είχε κριθεί από την δική μας Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ως ε, σχετικά άτολμη περιορισμένη και ελάχιστα φιλόδοξη πρόταση. Εμείς δώσαμε μάχη. Παλέψαμε με νύχια και με δόντια. Και προσπαθήσαμε να καθιερώσουμε αυτή την ισότητα ανδρών και γυναικών. Ταχθήκαμε υπέρ της ε, συμφιλίωσης της οικογενειακής ε, και επαγγελματικής ζωής. Γι' αυτό και οι πουδενοί δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με την ε, αφαίρεση από την οδηγία αυτή της νομικής βάσης, το άρθρο 141 της συνθήκης ως νομικής βάσης. Οπότε, στόχος της δικής μας Επιτροπής ισότητα των ε, Φίλων και Δικαιωμάτων της Γυναίκας είναι να συνεχίσουμε τη μάχη μας για την αποκατάσταση αυτής της ισότητας και για το συνδυασμό του οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που αφορούν το ωράριο εργασίας, την, τις, μη τυπικές, τις ατυπικές φόρμες εργασίας. Και αυτά δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Γιατί κάποια τυπικά και παρατεταμένα ωράρια μπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία των γυναικών. Οπότε οι τροπολογίες που λένε ότι αν η γυναίκα δεν το επιθυμεί, δεν θα πρέπει να υποχρεώνεται ούτε σε βραδινή βάρδια, ούτε σε υπερορίες. Αλλά άλλο ισχύει για την εργασία την Κυριακή της Αργίας σε ορισμένα επαγγέλματα. Δηλαδή θα πρέπει εμείς να συμβάλλουμε στη διακριτική μεταχείριση βάρος των γυναικών επειδή δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση ή επειδή δεν έχουν την ίδια ικανότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ε, μίας δουλειάς όπως οι άνδρες. να εργάζεται κανείς τη μέρα Κυριακές ή Αργίες και να εργάζεται σε νυχτερινή βάρδια ή να κάνει παρατεταμένες υπερορίες. Δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία οι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία και το μεγαλύτερα προσκόμματα στην επίτευξη συμφωνίας αφορούν το θέμα της άδειας πατρότητας. Και θα ήθελα να ζητήσω τη βοήθεια των διερμηνέων. Γιατί άλλο άδεια πατρότητας και άλλο γονική άδεια. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την άδεια πατρότητας με τη γονική άδεια. Η γονική άδεια ισχύει και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Η άδεια πατρότητας αφορά μόνο τον πατέρα, τον άνδρα. Όπως η άδεια μετρότητας αφορά μόνο τη μητέρα, τη γυναίκα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η διάκριση, αυτός ο διαχωρισμός και αυτή η διευκρίνηση. Και σε καμία περίπτωση στις τροπολογίες μας δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε τη γονική άδεια με την άδεια πατρότητας. Επιχειρηματολογώντας ότι ήδη υπάρχει πρόταση τη γονική άδεια, ότι ήδη έγιναν διαπραγματεύσει με του κοινωνικού εταίρου για τη γονική άδεια, άρα δεν χρειαζόμαστε άδεια πατρότητα. Επαναλαμβάνω, άλλο γονική άδεια, άλλο άδεια πατρότητα. Επιπλέον, το θέμα της γονικής άδειας όντως συμφωνήθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους και όντως ε, αποτελεί τμήμα μιας άλλης οδηγίας. Είναι όμως άνευ αποδοχών η γονική άδεια. Δεν αμείβεται η γονική άδεια. Οπότε και η αξία της είναι πολύ περιορισμένη και η χρήση της θα είναι περιορισμένη γιατί δεν θα πρέπει οι οικογένειες επιλέγοντας τη γονική άδεια να βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική θέση ή να έρχονται σε δινή οικονομική κατάσταση επειδή αποφασίζουν να αυξήσουν τα μέλη της οικογένειάς τους. Το αντίθετο χρειάζονται συμπλήρωμα. Από τη στιγμή που θα έχουν περισσότερα οικογενειακά βάρη, περισσότερα ε, παιδιά, πρέπει να έχουν και κάποιο βοήθημα. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, η νομοθεσία μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο τις τρεις άδειες. Την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια και ευελπιστώ ότι στο μέλλον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι αυτός ο σωστός δρόμος, δηλαδή μια κοινή αντιμετώπιση των τριών ειδών άδεια. Θα πρέπει να γίνει ε, μια αντιστοιχία των τριών ε, ειδών άδεια και να συμπεριλαμβάνονται και οι τρει σε μια ενιαία οδηγία όπως συμβαίνει στην Ισπανία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία που τη χάνουν ίση μεταχείριση στα τρία αυτά είδη άδεια. Πάντως, η άδεια πατρότητας ήδη υπάρχει στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών. Υπάρχει ήδη στην εθνική νομοθεσία. Γι' αυτό και πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν είμαστε πρόθυμοι να προσαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία στις εθνικές νομοθεσίες, σε μέτρα που ήδη υπάρχουν στι εθνικέ ένωμε τάξει και κυρίω να την προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή που μα ζητάει να συνδυάσουμε την άδεια μητρότητα με την άδεια πατρότητα. Γιατί και οι δύο άδειε είναι οι δύο όψει του ίδιου νομίσματο. Το δικαίωμα στη μητρότητα το δικαίωμα στην πατρότητα και η δικαίωμα τη παρακολούθηση ε, τη ανατροφή των ε, παιδιών ισχύει και για του άνδρε και για τι γυναίκε. Γιατί να διαφοροποιούμε λοιπόν τις δύο άδειε. Και από ενοιολογική άποψη, αλλά και από άποψη τη σύγχρονη θεώρηση του ρόλου του ανδρό στην κοινωνία και των ευθυνών που φέρει στον οικογενειακό κύκλο, όλα αυτά τα επιχειρήματα συνηγορούν υπέρ της συμπερίληψη στην οδηγία αυτή για την άδεια μητρότητα και την άδεια πατρότητας. Και ολοκληρώνω με το σχόλιο ότι ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, ότι όλοι θα συμβάλλουμε στην ευόδοση αυτής της πρότασης και στη βελτίωση αυτής της οδηγίας και τον εξυγχρονισμό της, προκειμένου να γίνει μια σύγχρονη οδηγία που θα είναι στραμμένη προς το μέλλον. Δεν μπορούμε να νομοθετούμε μόνο έχοντας υπόψη το παρόν. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο το σήμερα. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε και το αύριο και το μέλλον. Ήδη η παρούσα οδηγία ισχύει εδώ και 17 χρόνια. Η επόμενη οδηγία, η αναθεωρημένη οδηγία, θα ισχύσει για άλλα 10-20 χρόνια. Οπότε θα πρέπει να έχουμε υπόψη και το μέλλον. Θα πρέπει να είμαστε διορατικοί στην υποβολή των προτάσεών μας και να υιοθετήσουμε πιο μακρόπνοες προτάσεις. Σας ευχαριστώ Ευχαριστώ για τη συνεργασία και είμαι βεβαία ότι με τη συνεργασία θα καταφέρουμε καλή συμφωνία που θα δώσει κύρος και έγκλη και σε εμά και στο Κοινοβούλιο και κυρίως στις ευρωπαϊκές οικογένειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Εστρέλα ή κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Είναι ενδιαφέρον νομίζω. Το ότι ακούστηκε και η Επιτροπή και οι στατιστικές που μας ε, έχουν υποβληθεί που δείχνουν ότι άνδρες και γυναίκες ε, λίγο πολύ κερδίζουν το ίδιο μέχρι την ώρα που φτιάχνουν οικογένεια. Γυναίκε με μικρά παιδιά κερδίζουν λιγότερα από ότι οι άντρε συναδελφοί του ή οι άντρε συναδελφοί του με μικρά παιδιά. Δηλαδή γίνεται, ε, ε, ε, διαιωνίζεται το πρότυπο ότι ο άντρα είναι αυτό που εξασφαλίζει το βιοπορισμό τη οικογένεια και το πρέπει να κερδίζει περισσότερο. Για να έχουμε λοιπόν την ισότητα στην αγορά εργασία, θα πρέπει να φροντίσουμε και για την ισότητα αυτή. Δύο εβδομάδε. ναι. Μπορεί να μην είναι μεγάλη αλλαγή, αλλά είναι μια αρχή. Είναι μια καλή αρχή και ένα καλό μήνυμα που αποστέλει η Ευρώπη. Εν προκειμένου λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι όντως ενδιαφέρον η πρώην Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διευθύντρια, το ότι ήρθε η Γενική Διευθύντρια, πρώην Γενική Διευθύντρια στην Επιτροπή. Ήταν για πολλά χρόνια Γενική Διευθύντρια στην Επιτροπή, έχτισε την σταδιοδρομία της η κυρία Οντζίλ Κόντα. Και τι μας είπε. Ότι σε μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να διατυπώνονται νομοθετικές διατάξεις. Αυτό που χαρακτηρίζει όμως και ξεχωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πάντα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ότι πάντα έχει τις καλύτερες διατάξεις και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση έχει εκδώσει τις νομοθετικές διατάξεις πριν από τα ίδια τα κράτη-μέλη, τα τραβάει προς τα μπρος δηλαδή. Τώρα όμως η κατάσταση έχει αλλάξει, γιατί 15 κράτη-μέλη προβλέπουν δύο εβδομάδες ε, άδεια για τους ε, πατέρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο καλύτερα, χωλαίνει για να προλάβει τα, την προοδευτικότερη νομοθεσία στο θέμα αυτών των κρατών μελών. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω την εισηγήτρια την ε, άδεια πατρότητας υποχρεωτικά μέσα στην νομοθεσία. Ευχαριστούμε κυρία Λούκας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την κυρία Εστρέλα. Ήταν πολύ καλή η έκθεσή τη. Εξαίρετη συνεργασία κατά την προετοιμασία τη έκθεση. Πολύ καλή η προσέγγιση τη. Και ευχαριστώ ιδιαίτερω, συμφωνώ ιδιαίτερω με τη γραμμή την οποία υιοθέτησε και η ίδια και η κυρία Τόμψεν που μόλι ε, μίλησε. Δύο τροπολογίε μόνο έχουν καταθέσει οι πράσινοι. Η πρώτη αφορά την ε, παράταση του χρόνου της μητρότητας στις 24 εβδομάδες σε πολλά κράτη-μέλη, από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν 18 εβδομάδες αδιαμετρόπιτας. Φυσικά τις 20 εβδομάδες ε, τις οποίες δάει η κυρία Εστρέλα είναι σωστό, η σωστή κατεύθυνση. Αλλά εμείς ε, επιδιώκοντας καλύτερες συνθήκες ε, για τις γυναίκες και οι συμμεταχείρε, συζητούμε 24 εβδομάδες και γι' αυτό επιμένουμε ιδιαίτερα ότι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της άδεια πατρότητας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα θα ήθελα να την περιλάβει η έκθεση και ξέρω ότι είχαμε την παραθέση και στο παρελθόν, αλλά η πλειοψηφία των μελών της ομάδας μας, της Επιτροπής μας, ε, τίνει προς τη συμπερίληψη και της άδειας πατρότητας στην έκθεση. Ξέρω ότι πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει με μεγάλα λόγια για την πρόοδο αυτή, στην δυνατότητα για την άδεια πατρότητας κτλ. Αλλά δεν έχει κάνει πολλά πράγματα και το να συμπεριλάβουμε το αίτημα αυτό για δύο εβδομάδες άδειας πατρότητας μέσα στην έκθεση ήταν ένα τεράστιο άλμα που θα μας έφερνε και πιο κοντά στους στόχους μας. Επίσης, απαραίτητο είναι να είναι και υποχρεωτική αλλά και αμοιβόμενη η ε, μεταποδοχών, δηλαδή άδεια πατρότητας, γιατί εάν δεν είναι υποχρεωτική, αν είναι μόνο ε, προαιρετική, πολλοί είναι εκείνοι θα δεν θα την χρησιμοποιούν και πάνω απ' όλα αν είναι άνευ αποδοχών, ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ την κυρία Εστρέλα. Πολλούς μήνες συζητούμε το θέμα αυτό όπως γνωρίζετε. Οι πράσινοι έχουν υποστηρίξει εν γέννη την έκθεση αυτή και ελπίζουμε να δούμε την ε, βέλτιστη εξέλιξη στην ε, έκθεση. Μάλιστα η κυρία Κλάστορ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Στρέλα. Οι πολυάριθμες τροπολογίες που έχουν κατευθεί δείχνουν ότι υπάρχουν ε, πολλές διαφορετικές τοποθετήσεις. Εγώ δεν διαγιγνώσκω την ε, ομοθυμία την οποία θέλει να διαπιστώσει η κυρία Λούκας. Ε, από τις παρατηρήσεις και της Επιτροπής και της Προεδρίας δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλει το Συμβούλιο στην υπόθεση αυτή πολύ καλά, έχει τον στόχο της προστασίας της μητρότητας, καλύτερη προστασία της μητρότητας, όλοι το θέλουμε, αλλά αποφασιστικά μέτρα δεν βλέπω πουθενά. Και κυρία Στρέλλα, δεν αντιλαμβάνουμε πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι η πατρότητα είναι διαφορετική υπόθεση από τη γονική άδεια. Δεν είναι ο άλλος γονιός ο πατέρας. Γιατί δεν είναι άδεια, ε, γονική άδεια. Οι γονείς είναι ο πατέρας και η μάνα, έτσι. Η μάνα ναι, χρειάζεται την άδεια μητρότητα, χρειάζεται και την προστασία αμέσω πριν και μετά από την ε, γέννα, από τον τοκετό. Άδεια τοκετού λοιπόν, πολύ καλά. Αλλά με τον τοκετό τι σχέση έχει ο πατέρα. Ο πατέρα την εποχή κατά την οποία αναρώνει η μητέρα ε, και αναπτύσσεται η σχέση με το παιδί κτλ. έχει την δυνατότητα να συμβάλλει, να συμπαρασταθεί στη μητέρα. Είναι ταυτόχρονα όμως ένας γονιός ο πατέρας, ο οποίος έχει το ρόλο του να παίξει ως γονιός και μόνο ως γονιός. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Για την κυρία Τόμψεν, η οποία βλέπω ότι θέλει να μην ε, ε, χωλένουμε πίσω από την ε, προοδευτικότερη από το μέσο όρο νομοθεσία της πατρίδας της πρέπει να πω ότι και για μένα ισχύει το ίδιο. Εμεί έχουμε την προστασία τη μητρότητα και έχουμε και τη δυνατότητα τη προστασία τη γονικής άδεια για τον πατέρα, αλλά με διαφορετική ρύθμιση. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να το λάβετε υπόψη αυτό ότι υπάρχουν διαφορετικέ σχέσει μεταξύ ε, των ρυθμίσεων των κρατών μελών και πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Για τη Γερμανία έχουμε άδεια μητρότητας. 14 εβδομάδες μόνο για τη μητέρα. Έχουμε γονική άδεια ένα χρόνο και δύο μήνες τους οποίου, οποίους μπορεί μόνο ο πατέρας να λάβει. Εάν δεν αξιοποιήσει αυτούς τους δύο μήνες, τους χάνει η οικογένεια. Εάν αποφασίσουν και οι δύο γονεί να πάνε να δουλέψουν, δεν μπορούν να τους αξιοποιήσουν. Και το βρίσκω καλό αυτό. Είναι μια καινούργια ρύθμιση στη Γερμανία. Το χρησιμοποιούν οι γονείς όλο και περισσότερο και δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει όλα αυτά να μπουν μέσα σε ένα καζάνι, να ανακατευτούν και μέσα από το καζάνι αυτό να βγει κάτι διαφορετικό από ό,τι σχέση τα κράτη-μέλη μας. Παρακαλώ λοιπόν θερμά την κυρία Εστρέλα αυτήν την τροπολογία ε, και της ε, κυρίας Νίμπλερ, του Τόμας Μαν και της υποφαινομένης την υπαρθμόν 23 να την κάνει δεκτή γιατί αυτή η τροπολογία σας στόχο έχει να δούμε με ένα διαφορετικό φως αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη επιμέρους για την άδεια το ή την αδιαμετρότητα και την γονική άδεια. Τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη εισαγάγει. Αυτά πρέπει να τα ε, αξιολογήσουμε και να τα διαφυλάξουμε. το, την καλή εθνική νομοθεσία πρέπει να τη διαφυλίξουμε. Γιατί αυτό είναι προς και των οικογενειών. Η ε, προστασία της μητέρας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είναι η προστασία προ και μετά τον τοκετό της μητέρας. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα το να μιλούμε για γονική άδεια, η οποία θα πρέπει να ε, προβλεφθεί και για τους ε, πατεράδες και για τις μητέρες. Γιατί τότε με αυτό το σύστημα μπορούμε να έχουμε ένα μια καλή λύση για τις οικογένειές μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ. Με εξέπληξε κάπως η τελευταία αυτή παρατήρηση. Γιατί αν όλα είναι τόσο φως φανάρι, γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ με τη συμφωνία. Αυτό το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και θα είχαμε καταφέρει να διεκπαιρώσουμε το θέμα αλλά την τελευταία στιγμή βρεθήκαμε μπροστά στο εμπόδιο που όρθωσαν το ΕΛΚ τους φιλελεύθερους. Να το ξανασυζητήσουμε, μην ξεχνούμε δηλαδή γιατί προσκρούσαμε σε αδιέξοδο και καλούμαστε σήμερα να ξανασυζητήσουμε το ίδιο θέμα. Τώρα ως προς την ουσία του προβλήματος, η κυρία Στρέλα το εξήγησε. Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα της ε, Λεχώνας, που της που μόλις ε, ε, γέννησε, είναι ένα θέμα το θέμα της ανάνυψης της σωματικής και εξασφάλιση των δικαιωμάτων ε, της γυναίκας. Και όπως είπε η κυρία Λούκας, εμείς προτείναμε αντί 20-24 εβδομάδες άδεια. Γιατί αυτό προτείνει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως ε, ελάχιστη περίοδο για την ε, σωματική ανάκαμψη της γυναίκας. Ένα εξάμεινο. Αυτό είναι θέμα δικαιώματος της γυναίκας. Να ανανύψει μετά τον τοκετό και να απολαύσει αυτό το δικαίωμα της μητρότητας. Και μετά είπαμε να προβλέψουμε και την άδεια πατρότητας, ώστε στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας σωματικής ανάμνησης να μπορεί να τύχει τη στήριξη του συζύγου, του πατρός ή ε, γυναίκα. όταν υπάρχει φυσικά, γιατί υπάρχουν και μονογονεϊκές οικογένειες. Πάντως είναι απόλυτα συμβατά και τα δύο δικαιώματα και του, της άδεια μητρότητας και της άδειας πατρότητας και μπορούν και να συμπίπτουν. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε όχι μόνο την ανάγκη, αλλά και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτής της άδεια πατρότητας. Και μάλιστα, από την τελευταία παρατήρηση, διαμόρφωσα την εντύπωση ότι όλοι συμφωνούμε με το θέμα αυτό. Οπότε, προς τι αυτές οι δυσκολίες στο Συμβούλιο και αυτό το διέξοδο και επιφυλάξεις. Χαίρομαι που από ενιολογική άποψη συμφωνούμε. Επιμένω όμως στο θεμελιώδη στοιχείο. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, η 43 για παράδειγμα, όπου πολύ συγκεκριμένα και πολύ κατηγορηματικά απαιτείται ελάχιστος όρο ε, δύο εβδομάδων. Ίσως ε, η αφησιμία γίνεται ότι δεν είναι υποχρεωτικέ. Εμείς ζητούμε αυτή η άδεια να είναι υποχρεωτική. Για να μην είναι ένα δικαίωμα, αλλά μία ανάγκη και μία υποχρέωση. Και παρόλο που θα αφήνουμε ένα περιθώριο ελιγμό στα κράτη-μέλη, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι τουλάχιστον αυτέ οι δύο εβδομάδε, γιατί άλλοι είναι πολύ πιο φιλόδοξοι και πολύ πιο απαιτητικοί, αλλά χάρη συμβαστική λύση, παρόλο που θεωρούμε ανυπαρκή τι δύο εβδομάδε, είμαστε διατεθειμένοι να συμφωνήσουμε σε αυτέ, αρκεί να είναι υποχρεωτικέ. Α είμαστε έντιμοι και ειλικρινεί. Και όταν συζητούμε το θέμα αυτό, να πούμε ότι εδώ θα πρέπει να κατοχυρώσουμε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της άδεια πατρότητας, όπως πολύ σωστά μας εξήγησε και η συγγήτρια. Ω συμπλήρωμα όμως της άδεια μητρότητας του δικαιώματος των γυναικών που γέννησαν, για να ανανύψουμε τα τοκετό με τη βοήθεια και του συντρόφου. Επίσης, η άδεια θα πρέπει να ξεκινά από την ημέρα του τοκετού γιατί θα είναι κρίμα να συρρυκνώνουμε αυτό το δικαίωμα και για την περίοδο πριν το δοκετό, για τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γιατί μία έγκυος γυναίκα, όσο έγκυος και αν είναι, όσο προχωρημένη και είναι η εγκυμοσύνη, έχει κάθε δικαίωμα και είναι απόλυτα ικανή να ασκεί το επάγγελμά τη. Τώρα, δεν θα πρέπει να συρρυκνώνουμε αυτό το δικαίωμα και να ε, θέτουμε το σημείο αφετηρίας του και πριν το τοκετό. Κατά τη γνώμη μου αυτό θα ήταν επικίνδυνο και η ομάδα μου είναι κατά. Θα πρέπει άδεια να ξεκινάει από την ημέρα του τοκετού. Και υπάρχουν και κάποια θέματα μετάφρασης. Σε ορισμένε περιπτώσεις η αγγλική μετάφραση, στην τροπολογία 2 για παράδειγμα, μιλάει για το συνδυασμό της εργασιακής ζωής, work life. Αυτό στα αγγλικά είναι πολύ ευρύ. Στα ισπανικά όμως, και προσοχή εδώ, αναφέρεται ο συνδυασμός του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για το συνδυασμό του οικογενειακού ή και του εργατικού βίου, του επαγγελματικού, αλλά τον συνδυασμό ή την ε, συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Είτε είναι οικογενειακός αυτός, είτε είναι προσωπικός, ιδιωτικός. Πάντως ε, το αυθεντικό είναι το αγγλικό πρωτότυπο και με αυτό θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και οι υπόλοιπε μεταφράσεις. Ευχαριστώ. Ε, Μάλιστα ευχαριστούμε. Η κυρία τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω ότι δεν επέβαλε απέκλεισμο το ΕΛΚ ε, ζητώντας αναπομπή του εγκριθέντος κειμένου. Ένα λεπτά και θα σας εξηγήσω ε, το κείμενο που είχε εγκριθεί στην Επιτροπή Γυναικών. Το κείμενο που είχαμε εγκρίνει εδώ ήταν εντελώς ε, ατελές και δεν έκανε, δεν έκανε για νομοθετικό κείμενο. Ήταν δε και μη εφαρμόσιμο. Σώσαμε το κοινοβούλιο, θα είχε γελιοποιηθεί το κοινοβούλιο αν τελικά είχε εγκριθεί η έκθεση. Τώρα όμως διαπιστώνουμε, όπως λέμε και στα γαλλικά, ότι ορισμένες φορές βοή εν τη ερήμο είναι κάποιες προσπάθειες που κάνουμε Αλλά η συγγήτρια τι έκανε, χειροτέρεψε το κείμενο. Είναι ακό, επικρατεί ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση ε, και δεν ε, καταλαβαίνουμε. Και ήδη το αρχικό κείμενο δεν έκανε για νομοθέτημα. Μην ε, ξεχνάτε ότι ακολουθούμε μια νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Δεν είναι έκθεση πρωτοβουλία όπου γράφουμε ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι και γράφουμε όλες τις ευχές μας και γράφουμε, σημειώνουμε ό,τι, ό,τι μας περνάει από το μυαλό. Οι εργοδότες και οι μισθωτοί πρέπει στην καθημερινή του ζωή να εφαρμόσουν ένα νομοθέτημα απλό και σαφές που στόχο έχει πραγματικά να προστατεύσει την μητρότητα. Αυτός είναι ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής. Μην ξεχνάτε δε ότι ήδη έχουμε δύο διαφορετικές νομικές πράξεις πρώτον για την προστασία της μητρότατης και δεύτερον για τη γονική άδεια Μόλις εγκρίναμε ένα κείμενο ώστε να αποδώσουμε νομική ε, γυρότητα ε, σε μια ε, πρόταση των κοινωνικών εταίρων για την γονική έδεια. Και τώρα τι κάνουμε, τι κάνετε μάλλον, μπλέκεστε τώρα σε αυτό το θέμα όπως μπλέκεστε και στην άδεια μητρότητας. Και τελικά το αποτέλεσμα θα είναι να μην είναι απασχολήσιμοι ούτε και οι άντρες μετά τις γυναίκες. Σας παραπέμπω σε κάποιες ε, τροπολογίες ε, και ε, στις διακοπές που είχα ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά φέρωσα πάρα πολύ χρόνο για να καταλάβω περί πρόκειται. Λοιπόν, δεν θα μπορούν να εργάζονται πλέον νύχτα οι πατεράδες εφόσον είναι κάτω του ενός έτους το παιδί τους. Καλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την απασχολησιμότητα των αντρών. Ζητάτε και πάλι οι σε, αναπαραγωγική ηλικία άντρες να έχουν την ίδια προστασία για την υγεία τους όπως και οι έγκες. Ευνούχους θα τους κάνετε για να μπορέσουν να δουλεύουν ας πούμε στα ορυχεία. Μα πείτε μου, καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η πρόταση. Δεν αμφισβητώ τις καλές προθέσεις, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, γιατί ε, ναι, ας πούμε όσοι είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, άντρες και γυναίκες, ε, ε λοιπόν να μην εργάζονται πια, να σταματήσουν. Πώ θα τα μεγαλώνουν τα παιδιά του, δεν ξέρουμε. Πρέπει να έχουν εκατομμύρια, έτσι. Ε, μάλλον, συγγνώμη, εκατομμύρια ε, ανθρώπων στην Ευρώπη δεν μπορούν να δουλέψουν ενώ θέλουν. Οπότε μην τα χειροτερεύουμε τα πράγματα καθιστώντα μία απασχολήσουμε του άντρε και μία απασχολήσουμε στις γυναίκε με τέτοιε τροπολογίε Καλοπροαίρετε είναι. Δεν λέω, αλλά περισκεπτέ. Τώρα αν θέλετε να είναι μέσα σε μια ενιαία νομική πράξη η προστασία της μητρότητας, η γονική άδεια και η άδεια πατρότητας, ε, ζητήστε το. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει αναπέμψτε την πρόταση στην Επιτροπή και ζητήστε το. γιατί εμείς με αυτές τις τροπολογίες ε, δεν δυνάμεθα να εκπονήσουμε νομικό κείμενο που ακόμη, ακόμη και αν εγκριθεί στην Ολομέλεια γιατί πλέον δεν είναι πολιτικός ορθό ε, να ε, αντιτάσσεται κανείς σε όλες αυτές τις τροπολογίες ε, που είναι τρελές, αντικρουόμενες. Δεν αρμόζει αυτό σε ένα νομοθετικό κείμενο που καλούνται να εφαρμόσουν και επιχειρήσεις και εργοδότες και οι μισθωτοί. Λοιπόν, ξαναλέω, ζητήστε καινούριο κείμενο, καινούρια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι μια νομική πράξη που να καλύπτει ταυτόχρονα και την προστασία της μητρότητας και τη γονική άδεια και την άδεια των ε, πατρότητας επανειλημμένα έχει πει η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξάλλου ότι επιθυμεί ε, με μονομένες νομικές πράξεις, θέμα, δηλαδή για την προστασία διαφορετικών θεμάτων. Ωραία. Ε, ας ζητήσουμε πράξη για την προστασία της ε, μητρότητας. Οι κοινωνικοί εταίροι δε τώρα συζητούν νέες πρωτοβουλίες. Όπως που ανέλαβαν την πρωτοβουλία για τη γονική άδεια, τώρα λοιπόν συζητούν μια αντίστοιχη πρωτοβουλία που θα μπορούσε να γίνει νομικός δεσμευτική, όπως μια οδηγία, ε, παραδείγματος χάρη, για την άδεια πατρότητα. Σας περιμένουμε. Αν θέλετε τώρα να, να, να σπεύσετε, εστιάστε την προσοχή σας ε, στην προστασία της μητρότητας που έχει την καθοριστική σημασία, τη ζωτική σημασία, αν πραγματικά θέλετε να προστατεύσετε τη μητέρα και το παιδί. Τώρα, αν ε, ε, θέλετε ένα συνονθήλευμα, τίποτα δεν θα καταφέρουμε. Γιατί ακόμη και αν εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση και περιέχει όλες αυτές τις προτάσεις που άσχετες είναι με την προστασία της μητέρας και του παιδιού, ε, λοιπόν θα αποτύχουμε παταγωδό στη δεύτερη ανάγνωση ε, και θα επιβραδυνθεί η ε, βελτίωση της προστασίας της ε, μητρότητας. Ξέρετε, θα σταματήσω εδώ γιατί δύο ώρες θα μίλαγα άμα μου ζητούσατε να σχολιάσω όλες αυτές τις γελίες προτάσεις που βλέπουμε μέσα στο κείμενο και στις τροπολογίες. Διακόπτει η Πρόεδρος. Συγγνώμη κυρία Λούλινγκ, συνοψίστε και κλείστε γιατί δεν έχουμε και τόσο πολύ χρόνο, μάλιστα, Πρόεδρε. Ε, δεν σας αρέσει να τα ακούτε, γι' αυτό θέλετε να με διακόψετε. Ξέρετε, εδώ επικρατεί δημοκρατία και έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε, γιατί θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος και ακριβώς γι' αυτό έχουμε το θάρρος να ισχυριστούμε ότι αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Κάντε εσείς ό,τι θέλετε τώρα βέβαια, αλλά εγώ σας υπόσχομαι ότι θα αποτύχετε και πάλι. Προεδρο. ευχαριστώ. Κυρία Λούλινγκ, σύσσωμη σα ακούσαμε με προσοχή. Έχουμε όμως άλλο ένα 20 λεπτό και μετά τελειώνει η συνεδρίαση και έχουμε ένα μακρύτατο κατάλογο ομιλητών. Όλους τους ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα. Η κυρία Κορνέλισεν και μετά η κυρία Ζαμπόσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Λούλινγκ. Μερικές φορές γελιοποιείται το Κοινοβούλιο όπως και η Επιτροπή μας. Αλλά οι λόγοι δεν, είναι, δεν εντοπίζονται στην έκθεση αυτή. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της γελιοποίησης, του εξευτελισμού. Εγώ είμαι υπέρ της γραμμής που ακολουθεί η κυρία Στρέλα. Θα ήθελα όμως να δούμε λίγο την ευρύτερη εικόνα της κατάστασης. Τα επόμενα δέκα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο γυράσκοντα πληθυσμό και θα χρειαστούμε την συνδρομή στην αγορά εργασίας, την παρουσία στην αγορά εργασίας κάθε ικανού άνδρα και γυναίκας. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και παιδιά να κάνουμε και οι γυναίκες θα πρέπει να είναι σε θέσεις που λαμβάνουν αποφάσεις και οι γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι θα πρέπει οι πάντες να έχουν τη δυνατότητα και να εργάζονται και να μεριμνούν για τα μέλη της οικογένειάς τους, αλλά ταυτόχρονα αυτό να γίνεται και ελκυστικό και ιδιαίτερος για τις γυναίκες. Και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και ένα ελκυστικό πακέτο για την άδεια. Είναι ελκυστικό για μια γυναίκα να έχει επαρκή ε, άδεια την ώρα που κάνει ένα παιδί, αμέσω μόλι κάνει ένα παιδί, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αποχωρήσει από τη θέση εργασία τη. Τα 20, 20 εβδομάδε προτείνει η κυρία Στρέλα είναι το ε, απολύτω ελάχιστο. Η δική μου εμπειρία ω εργοδότη από την ε, πρόσφατη μου σταδιοδρομία είναι ότι όταν είναι πολύ σύντομη η άδεια, ο, ο ενδιαφερόμενο ε, αξιοποιεί την ετήσια άδειά του. Ή και όταν αργότερα ε, χρειαστεί την άδεια, την αιτήσια για να πάει διακοπές, αναγκάζεται να πάρει άδεια ασθενεία. Ή αμέσω μετά την άδεια μητρότητα χρησιμοποιεί την άδεια ασθενεία εφόσον δεν έχει άλλη λύση. Θα χρειαστούν λοιπόν ίσω και θα ήταν υπεροστόφελο και του εργοδότη να έχουμε καλύτερη ε, μακρύτερη άδεια μητρότητα. Είναι πολύ πιο εύκολο να αντικατασταθεί μια γυναίκα στην άδεια μητρότητα με μια-δύο εβδομάδε παραπάνω, γιατί μέχρι να βάλουμε κάποιον μέσα στη δουλειά, να του εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνει, ε, έχουμε χάσει πολύ χρόνο. Για τον εργοδότη, λοιπόν, δεν είναι μεγάλη επιβάρυνση και ίσω να το θεωρήσει και ευπρόσδεκτο μέτρο. Επίση, απαραίτητο είναι να δώσουμε άδεια με πλήρε αποδοχές στον πατέρα Εάν δεν είναι πλήρε οι αποδοχέ, δεν θα πάρει την άδεια, γιατί πολλέ είναι οι οικογένειε που εξαρτώνται για την επιβίωσή του από την άδεια του πατέρα. Και πρέπει να είναι παρόν ο πατέρα τι πρώτε δύο εβδομάδε τη ζωή του παιδιού. Η Γερμανίδα συνάδελφο είπε ότι αργότερα μπορεί να βοηθήσει ο πατέρα. Όχι λοιπόν, τι δύο πρώτε εβδομάδε θα μάθει να αλλάζει το πάμπερ, τι δύο πρώτε εβδομάδε θα, βάλει, θα μάθει να κάνει το μωρό του μπάνιο ή να το βάζει στο κρεβάτι. Και μόνο τι δύο πρώτε αυτέ εβδομάδε μπορεί να αναπτυχθεί η ρουτίνα στην οικογένεια που θα βοηθήσει και τον πατέρα να συμμετάσχει σε όλη αυτή τη φροντίδα για το παιδί. Γιατί διαφορετικά έχει ξεκινήσει μια ρουτίνα και ο πατέρα δεν μπορεί να συμμετάσχει ούτε καν βρίσκει τρόπο να μπει μέσα αυτή τη ζωή τη οικογένεια. Πολλοί ήταν οι άντρε με του οποίου εγώ έχω συνομιλήσει και μου είπαν ότι θα ήθελαν υποχρεωτική την ε, άδεια πατρότητα. Βρίσκουν ει βάρο του διάκριση το γεγονό ότι δεν του επιτρέπεται να ε, συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση τη ζωή του παιδιού του, στην πρώιμη φάση. Και λυπούμε που το ΕΛΚ δεν θέλει να συμπεριληφθεί η άδεια πατρότητα στη συγκεκριμένη οδηγία. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Στρέλα ότι θα πρέπει να είναι ένα και ενιαίο πακέτο, μια ενιαία δέσμη μέτρων αυτή η άδεια, η άδεια μητρότητα πρόταση άδεια πατρότητας και η γονική. Ε, εν τέλει, ωστόσο, εάν καταστεί η προαιρετική αυτή η άδεια πατρότητας, θα πρέπει να δούμε τι συνέπειες θα έχει αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, όπως λέει η κυρία Λούλινγκ, ε, μια χωριστή οδηγία για την γονική άδεια. Πολύ καλά, αλλά ακούσαμε και τον κύριο Ανδρός και την κυρία Ρέντινγκ και δεν φάνηκε να έχουν τέτοιες προθέσεις. όλοι εκεί ήμασταν, τα ακούσαμε, τα ίδια λόγια ακούσαμε όλοι. Δυστυχώς, ξέρουμε όλοι ότι δεν έχουμε το δικαίωμα της πρωτοβουλίας, δεν μπορούμε να προκαλέσουμε εμείς σύνταξη νομοθετικού κειμένου και γι' αυτό προτείνω όσοι είναι υπέρ της γονικής, της άδειας πατρότητας, με οποιοδήποτε μορφή και αν θέλουμε να υπάρχει αυτή, να υπερψηφίσουν τη σχετική πρόταση. Η ε, κυρία Σαμπόσκά, και σας ενημερώνω ότι έχουμε άλλους έξι ομιλήτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα είπαν οι προλαλήσαντες, θα περιοριστώ σε κανένα δυο σχόλια. Όταν ε, πρωτοξεκίνησε αυτή η συζήτηση για την οδηγία, το γεγονός ότι Συμπεριλάβουμε στη συζήτηση και το θέμα της άδεια πατρότητας είναι σαν να ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας. Και τώρα δεν μπορούμε να διεκπαιρώσουμε τη συζήτηση. Είναι κρίμα, αλλά ούτε και η σημερινή συζήτηση δεν διαφέρει από την συζήτηση της προηγούμενης άνοιξης. Η βασική αρχή είναι να εμείνουμε στον τίτλο αυτής της οδηγίας και να μην επεκταθούμε τα... δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε νέα κεφάλαια και να συμπεριλάβουμε νέα θέματα στη συζήτηση. Να επικεντρωθούμε στις γυναίκες και στην άδεια μητρότητας. Αυτό είναι το πεδίο εφαρμογή οδηγία. Και τις δύο εβδομάδες κάναμε 14 για να βοηθήσουμε τις γυναίκες να συνηθίσουν στη νέα κατάσταση. Να εγκληματιστούν στον καινούριο τους ρόλο Νομίζω ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το Συμβούλιο, ούτε οι Προεδρίες, οι Σουηδικοί προηγουμένως, η Ισπανική τώρα, δεν έχουν αποκρισταλωμένη γνώμη για το περιεχόμενο της οδηγίας. Ακούσαμε τις προθέσεις της Ισπανίδας Υπουργού για το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας σε θέματα ισότητας, αλλά δεν μας φώτισε και όλα για το ποια είναι η σαφής γνώμη της Ισπανικής Προεδρίας. Φυσικά δίνουμε έμφαση και μας ενδιαφέρει η ισότητα και εγκρίναμε την έκθεση Ταραμπέλα, ακούσαμε για τα κριτήρια της Βαρκελόνης, ακούσαμε για τους στόχους της χιλιετίας και έγινε και λόγος για μερικούς τομείς. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η οδηγία αυτή δεν πρόκειται να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη. Θα είναι ανέφικτη η εφαρμογή της. Και διατρέχουμε το κίνδυνο να δημιουργηθούν ανισότητες και στους μισθούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό το φαινόμενο, το ζούμε εδώ και 50 χρόνια. Και θέσαμε και σχετική ερώτηση στην Υπουργό. Σίγουρα και οι άνδρες, οι πατεράδες μπορούν να μάθουν να φροντίζουν το, το νεογέννητο. Ακόμη και αν δεν βρεθούν στο σπίτι από την πρώτη μέρα της ζωής του. Μπορούν να εξοικειωθούν με τη ζωή του βρέφους. Δεν χρειάζεται να έχουν άδεια πατρότητας από την πρώτη μέρα μετά το τοκετό. Η κυρία Ορή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να διορθώσω ένα λάθος που υπόθηκε. Σε καμία περίπτωση οι φιλελεύθεροι δεν μπλοκάρισαν αυτή την οδηγία. Στην τελική ψηφοφορία υπευλήθη ένα εγγραφό με πολύ επίμαχες και αντιφατικές θέσεις ε, με αποτέλεσμα να έχουμε την τελική ψηφοφορία και το τελικό αποτέλεσμα που θυμάστε. Εμείς είμαστε υπέρ της ε, έγκρισης μιας τέτοιας οδηγίας και η φιλελεύθερη είναι υπέρ της επέκτασης της άδεια μητρότητα σε 20 εβδομάδες τουλάχιστον, όπως πρότεινε η κυρία Στρέλα. Επίση είμαστε υπέρ της συμπερίληψη της άδεια πατρότητα στην ίδια οδηγία. Τουλάχιστον ε, οι φιλελεύθεροι που είναι μέλη της Επιτροπής ε, για τα Δικαιώματα της Γυναίκας είναι υπέρ αυτής της ε, πρότασης. Βέβαια το κόμμα μας δεν έχει καταλήξει σε οριστική γνώμη. Αλλά κατά τη γνώμη μου και η άδεια μητρότητας και η άδεια πατρότητας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί να περιμένουμε άλλα δύο-τρία χρόνια για μια νέα οδηγία που θα παρτίζεται από λίγες μόνο διατάξεις που θα ρυθμίζουν το θέμα της άδειας πατρότητας αποκλειστικά. Ας την περιλάβουμε από τώρα στην οδηγία. Από νομική πάντως άποψη, η άδεια πατρότητας δεν είναι γονική άδεια. Η γονική άδεια είναι μία δυνατότητα επιλογής που δίνεται είτε στον ε, πατέρα είτε στη μητέρα. Τώρα έχουμε δύο ξεχωριστές δυνατότητες, μία επιλογή για, για τη μητέρα και μία επιλογή για τον πατέρα. Εγώ ως δικηγόρος δεν είμαι υπέρ της υποχρεωτικής ε, εφαρμογής τη άδεια πατρότητας. Είμαι υπέρ μια άδεια πατρότητας μεταποδοχών, αλλά να αφήνεται η διακριτική ευχέρεια στον ε, πατέρα να αποφασίζει αν τον ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα και να ασκήσει αυτή την άδεια για να έρθει σε επαφή με το βρέφος. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 50 χρόνια, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών. Και είναι κρίμα να φοβούμαστε ότι το Συμβούλιο δεν θα το υποστηρίξει. Εγώ εξελέγην από το λαό της Εστονίας και όχι από την εστονική κυβέρνηση. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Αν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α, να εκφράζει πραγματικά τη γνώμη των ψηφοφόρων, τη γνώμη του λαού, θα πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση προς το Συμβούλιο για να το μεταπίσουμε προς τη δική μας κατεύθυνση, γιατί αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Ε, η άδεια πατρότητας να είναι δικαίωμα του πατρός και να είναι μεταποδοχών. Όχι υποχρεωτικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απαγόρευση νυχτερινής εργασίας για τους πατέρες, ε, διαφωνώ με τις διατάξεις αυτές. Θα πρέπει να διαβάσουμε πολύ προσεκτικά την πρόταση. Ευχαριστούμε η κυρία Φιγκρέντο και η κυρία Μπάουερ. Μην ξεχνάτε το χρόνο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ακούστηκαν πολλά ήδη. Παρ' όλα αυτά θα επαναλάβω τρία πράγματα. Πρώτον, το δικαίωμα που έχουμε όλοι να υποβάλουμε τροπολογίες. Και το κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να αποποιείται το ρόλο του. Ποιος είναι αυτός? Να εισηγείται πράγματα για να αναβαθμίσει τις προτάσεις της Επιτροπής. Κοιτάξτε, αυτό επισύρει κάποια καθυστέρηση, αλλά νομοθετούμε για το μέλλον. Ακούσαμε διάφορα επιχειρήματα εδώ, εν πάση περιπτώσει, για να ε, υποστηρίξουμε τη θέση ότι η άδεια πατρότητας ε, προσωμιάζει την άδεια μητρότητας. Ε, προφανώς, εδώ στο Κοινοβούλιο συνήθως λένε όλοι ότι θέλουμε αύξηση γεννητικότητας και ανησυχούν όλοι από την έλλειψη παιδιών. Αλλά όταν περνάμε στην πράξη, στη δημιουργία όρων ώστε να αυξηθεί και η μητρότητα και η πατρότητα και ενίσχυση της γενετικότητας, Τελικά τι κάνουμε, καταλήγουμε σε τέτοιες ε, συζήτησεις όπως ε, η σημερινή. Και να δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που ακούσαμε από τους συναδέλφους. Γι' αυτό το λόγο ήρθε η στιγμή ανεξάρτητα από τη διάσταση απόψεων. Να κάνουμε, ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα. Η συνάδελφός μας, η κυρία Εστρέλα, υποχώρησε σε κάποια σημεία μέσα στην έκθεση. Και ε, η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση στην προηγούμενη θητεία. Δηλαδή, εγώ στροπολογίες επαναλαμβάνω ε, προτάσει που είχαν εγκριθεί στη, από την Επιτροπή μας ε, στην προηγούμενη θητεία και που δεν έχουν συμπεριληφθεί μέσα στην έκθεση κυρία Εστρέλα και ε, απευθύνομαι στην κυρία Λούλιν και σε άλλους. Δηλαδή, άλλαξε την έκθεση. Πολύ κυρία Εστρέλα και η απόδειξη είναι ότι εγώ προτείνω επανεισαγωγή σημείων της έκθεσης που είχε εγκριθεί εδώ στην Επιτροπή την προηγούμενη θητεία. Δεν ε, αληθεύει αυτό που είπε η κυρία Λούλινγκ ότι την άφησε άθικτη την έκθεση η κυρία Εστρέλα την άλλαξε. Εγώ ίδια ε, ε, υποβάλλει αυτές τις προτάσεις και καταδεικνύω έτσι ότι υπήρξαν ε, αλλαγές μέσα στην έκθεση και πιστεύω ότι πρέπει να επανεσύχθουν κάποιες διατάξεις για τους 24 μήνες, 24 εβδομάδες συγγνώμη, στην αρχή είχαμε προτείνει 22, μετά καταλήξαμε στο 20, νόμιζα ότι ήταν συνενετική λύση, ε, ε, αυτό είναι το ελάχιστο όριο στο οποίο επιμένω για την άδεια πατρότητας. Ε, φυσικά θέλουμε να την υπερασπιστούμε για όλα αυτά που ακούσαμε. Και εν γέννη συμφωνούμε με την έκθεση. Τονίζω όμως ότι έχουν αφαιρεθεί προτάσεις που κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ σημαντικές και γι' αυτό μπαίνουμε στις τροπολογίες μας. Ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στις συναδέλφους τη συζήτηση πριν από ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, όταν είδαμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε, η οποία υποσχόταν ότι μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2009, θα μας καταθέτε προτάσεις για την άδεια πατρότητας. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις για τρία διαφορετικά θέματα και πρέπει να υπενθυμίσουμε στις συναδέλφους ότι δεν έχει υποβληθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άδεια πατρότητας, γιατί η κυρία Εστρέλα συμπεριέλαβε στο πακέτο αυτό την υγεία μάλλον τι συμπεριέλαβε στο πακέτο περί υγείας και ασφάλειας του χώρου εργασία. Πρέπει να δούμε πώς θα υποβληθεί η πρόταση και πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι λύπηρο το γεγονός ότι ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε ολοκληρώσει την υπόθεση αυτή, περατώσει την υπόθεση αυτή, βρισκόμαστε τώρα ακόμη να συζητούμε τα ίδια πράγματα. οι πληροφορίες που μας ε, προσφέρει η κυρία Εστρέλα είναι σφαλμένες το ότι η γονική άδεια δεν αμείβεται. Δεν υπάρχει κράτος μέλος που να μην προσφέρει αμοιβή, ε, που να μην διατηρεί δηλαδή τις αποδοχές στην ε, γονική άδεια. Υπάρχει όμως η δυνατότητα της μη μεταφερόμενης γονικής άδειας για τον πατέρα. Non-transferable. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ είναι δυνατόν ένα χρόνο να μιλάμε για το ίδιο πράγμα και ακόμα να είμαστε στη διάθεση και κάνουμε σημειωτών. Είχαμε το ίδιο πρόβλημα και με την οδηγία για το χρόνο εργασία και πρέπει επιτέλου να προχωρήσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να προχωρήσουμε. Υπάρχουν πολλοί ακόμη που έχουν ζητήσει το λόγο. Δυστυχώ όμω ο χρόνο μα εξαντλήθηκε. Πρέπει ωστόσο να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για την ε, συζήτηση. Ήταν πολύ ζωντανή. Σας ευχαριστώ. Ε, οι διερμηνείς μας έχουν διαθέσει μερικά λεπτά ακόμη, ώστε να επιτρέψουμε στην κυρία Εστρέλα να ε, μιλήσει για να κλείσουμε το, το θέμα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά για την συνεισφορά σε αυτή την πλούσια, ζωηρή, σφοδρή και συμμετοχική συζήτηση και ευχαριστώ και τους διερμηνείς που μας παραχώρησαν ε, λίγο ακόμη χρόνο για την ολοκλήρωση της συζήτησης. Για να επιτευχθούν συμφωνίες χρειάζεται κάποια διαλλακτικότητα και μία διάθεση προόδου και από τους μεν και από τους δε. Αυτή την προσπάθεια έκανα εγώ για να συμφιλιώσω τις διστάμενες απόψεις και έκανα πολλές υποχωρήσεις σε σχέση με την αρχική μου θέση. Και μάλιστα διαπίστωσα ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν προχώρησε καθόλου στη συζήτησή του. Ήταν ανένδοτο, ανυποχώρητο και καθόλου διαλλακτικό όπω οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε και αυτό θα ήθελα να το τονίσω. Θα ήθελα να θέσω δύο-τρει ερωτήσει ε, για να τι σκεφτείτε. Πρώτον, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσθέσει το άρθρο 141. Και μία υποερώτηση. Για ποιο λόγο πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία θα πρέπει να απασχολήσει ως κατ' αρμόδια την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και όχι την ε, Επιτροπή Απασχόλησης, γιατί η νομική βάση είναι το άρθρο 141. Μία άλλη ερώτηση που σας υποβάλλω ως για σκέψη, μετά από την ερώτηση της κυρίας Μπάουερ, είναι ποια είναι η αμοιβή που προβλέπετε για τη γονική άδεια μετά από συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Ποιο είναι το ύψος αυτών των αποδοχών. Υπάρχει άνδρας που είναι διατεθειμένος να στερηθεί το μισθό του για να παραμείνει στο σπίτι και να αναλάβει τη μέρη με των παιδιών ή να συμμετέχει στην ανατροφή και τη φροντίδα των παιδιών. Ποιος άντρας θα το κάνει αυτό. Επίσης, εμείς ε, με συνέπεια και αποφασιστικότητα προσπαθήσαμε να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε μορφή διακριτικής μεταχείρισης. Αλλά αν προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε τους άνδρες από τις οικογενειακές τους ευθύνες, προς αυτούς επιβάλλουμε διακριτική μεταχείριση. Είναι σαν να τους στερούμε το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τη γέννηση και την ανάπτυξη των παιδιών τους. Και οι άνδρες έχουν ίσα δικαιώματα με, του, με, τις, με τις γυναίκες. Ειδικά στην πρώτη φάση μετά το τοκετό που χρειάζεται η γυναίκα για να ανανύψει σωματικά. Και σίγουρα οι οικογενειακέ ευθύνε στην περίπτωση αυτή και μέρη με των παιδιών μπορεί να καταμεριστεί ισότιμα μεταξύ των ανδρών και γυναικών, μεταξύ των πατεράδων και των μητεράδων. Και αυτό είναι απαραίτητο για την οικογενειακή ισορροπία. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και διάφορα, ότι λεφτά υπάρχουν για όλου ή ότι δεν έχουμε κονδύλια για τα ουσιώδη. Αλλά θα πρέπει να βρούμε πόρου για να αποκαταστήσουμε μια αρμονία στον οικογενειακό βίο. Και αυτοί που είναι υπέρμαχοι της οικογένειας ε, θα πρέπει να είναι συνεπείς με τις αρχές τους και να φροντίσουν να βρουν κάποιους πόρους ε, γιατί δεν θα πρέπει να προβλέπουμε μόνο για τα κοινωνικά θέματα και για τα φάρμακα ε, πόρους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην οικογένεια και ψυχολογικά και πολλές φορές ε, οδηγούν σε ένα ιατρείο, σε μια ιατρική συμβουλή ή σε λήψη φαρμάκων. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 122 της κυρίας Γκαρσία Πέρες. Η οδηγία αυτή, η τροπολογία συγγνώμη αυτή είναι πολύ σημαντική. Και ίσως μας βοηθήσει να υπερκεράσουμε πολλά προβλήματα. Η κυρία Γκαρσία Πέρες είναι λίγο πιο φιλόδοξη από την τροπολογία 123 της κυρίας Κλάς έχει ένα τμήμα που είναι ταυτόσιμο με την 123, αλλά προτιμώ την 122 τροπολογία από την 123. Διαβάστε την προσεκτικά λοιπόν την τροπολογία 122, προβληματιστείτε. Πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τα διέξοδο και να υπερβούμε κάποιες δυσκολίες. Επειδή λοιπόν ο χρόνος μας πιέζει και τον εξαντλήσαμε, θα σταματήσω εδώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Εστρέλα, ευχαριστούμε όλους του συναδέλφου εργαστήκαμε πολύ εντατικά. Ε, αμοιβαίο σεβασμό παρακαλώ να δείξετε και να σέβεστε τις διστάμενες απόψεις. Οι συζητήσεις μας εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι σημαντικό να ακούμε οι μεν επιχειρήματα των δε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Ιστραέλα, ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το απόγευμα και η πρόταση ευγενικά ευχαριστεί και τους διερμηνείς που έδωσαν κάποια έξτρα λεπτά. Ευχαριστούμε και εμείς. Αύριο στις 9 οι συντονιστές θα συνεδριάσουμε. Ευχαριστώ.